ε, ήρθατε ε, κύριε Πρόεδρε Ράινα, αγαπητοί Ε, Έχουμε αυτή την ε, συνεδρίαση της ε, Διακοινοβουλευτική Συνέλευσης η οποία επικεντρώνεται στο θέμα πώς είναι δυνατόν να γίνει κανείς παγκόσμιος ηγέτης στον αγώνα της κλιματική αλλαγής. Αυτό είναι το θέμα το οποίο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ε, επισήμαναν στα κράτη-μέλη στην αρχή της ε, κοινοβουλευτικής θητείας για να αναλάβουν τα κράτη-μέλη περισσότερες ε, πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να τροποποιήσουν το μοντέλο ανάπτυξης. Ξεκινάμε λοιπόν από κάτι που πλέον όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο και αναγκαίο, δηλαδή να διασωθεί ο, πλανήτης. Και όλοι θέλουν να αγωνιστούν για την κλιματική αλλαγή, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατορθώσουν, να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις και να μπορέσουν να επερασπιστούν το δικό τους το κοινωνικό μοντέλο. Η κοινοβουλευτική αυτή εβδομάδα ε, μπορεί να θεωρεί ότι είναι πολύ επιτυχημένη όσον αφορά τη συμμετοχή. Πλέον αυτή η κοινοβουλευτική εβδομάδα είναι κάτι το απολύτω απαραίτητο στο ε, χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε την Κροατική Προεδρία για την πρωτοβουλία που ανέλαβε για τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο διοργάνωσε την εβδομάδα. Ε, οι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ε, οικονομικές πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις που θα κληθούμε να λάβουμε έχοντας ε, κατά νου την απαραίτητη ευρωπαϊκή διάσταση. Οι αποφάσεις μας λοιπόν έχουν συνέπειες για τους εταίρους μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γίνεται κοινωνός των δικών μας των απόψεων αλλά και των απόψεων των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πέτεινε την ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα Εθνικά Κοινοβούλια και αυτά όλα με στόχο να δείξει τις πράξεις της πρωτοβουλίας κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο Επίτροπος Γνωρίζω ότι μας έχει καλέσει σε διαβουλεύσεις, διαβουλεύσεις οι οποίες θα έχουν ως στόχο να απλουστευτεί το, πλαίσιο της, το υπάρχον πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης. Γιατί ε, πρόκειται για τους κανόνες του προϋπολογισμού που έχουν εγκριθεί στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Γνωρίζω λοιπόν ότι είχατε ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος. Ε, αυτή η ανταλλαγή απόψεων απόψεων ευωδόθηκε και το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο, σε αυτό το εξάμεινο εντάχθηκαν και στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόρθωσε να εισακούσει την άποψη των Ευρωπαίων πολιτών που ανησυχούν ιδιαίτερα για τα ε, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Η πρόοδος και η ανάπτυξη που έχουν επιτευχθεί δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν και τα μηνύματα των Ευρωπαίων Ευρωπαίων πολιτών, κυρίως αυτών που εκπέμπθηκαν στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής εβδομάδας. Η δική μας λοιπόν η συνεργασία, η συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια για μας είναι εκ των όνου κάνευ και απολύτως απαραίτητη. Έχοντας ε, δει τα θέματα που τίθενται νομίζω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε συμβιβασμούς προς όφελος όλων. Και όταν λοιπόν μιλάμε για ευρωπαϊκούς θεσμούς, αναφορά δεν γίνεται μόνο στους θεσμούς των Βρυξελών. Όλοι καλούμεθα να προσφέρουμε και εμείς ε, το δικό μας το κομματάκι στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και βεβαίως τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτή τη συνεισφορά. Αυτό που με ανησυχεί σήμερα είναι ο κίνδυνος της κατάτμισης του ευρωπαϊκού χώρου. Ένας κίνδυνος ε, που ε, αφορά την εθνική ταυτότητα η οποία θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να χάσουμε το, από τα μάτια μας την κοινή ευρωπαϊκή μοίρα. Γιατί πολλοί επισημαίνουν το θέμα της ε, κυριαρχίας που είναι σημαντική για όλους μας αλλά και της αλληλεγγύης ε, που είναι σημαντική για όλους και απαραίτητη εξάλλου. Αυτή λοιπόν η κατάτμιση, ο κατατεμαχισμός, αυτά τα διαπιστώνουμε στην ε, κοινή γνώμη. Βλέπουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τελείως διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι οποίοι εποφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση και υπάρχουν και άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι δυστυχώς αισθάνονται ότι στερούνται αυτές τις ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν η πολιτική κινητικότητα κατά την άποψή μας ε, μπορεί να θεωρηθεί ως μια πολιτική χήμερα. Υπάρχουν ε, αδυναμίες, προβλήματα ε, στα κράτη-μέλη, ε, στο βορρά και στο νότο της Ευρώπης, στην Ανατολή. Το, η ευρωπαϊκή διάσταση και ο ευρωπαϊκός βηματισμός σημαίνει ότι δυστυχώς υπάρχει και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσά μας. Απόσταση ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, το Βορρά και το Νότο, το κέντρο και τις περιφέρειες. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα όπου όλοι καλούμεθα να συνεισφέρουν ξέρουμε, ευρωπαϊκοί, εθνικοί θεσμοί. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα σημαίνει να αναζητήσουμε τρόπους έτσι ώστε να μειωθεί η απόσταση. Θα ήταν βέβαια πάρα πολύ ωραίο αν κάποια μέρα τα προβλήματα του Βορρά μπορούσαν να ε, εξεταστούν, να αντιμετωπιστούν από το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνικής γνώμης ως προβλήματα που αφορούν όλους. Και το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα προβλήματα του Νότου. Πολύ συχνά ο Νότος ε, ε, αντιμετωπίζει προβλήματα που διαχέονται και δημιουργείται ένταση. Άρα δηλαδή όλα αυτά τα ε, τα συνειδητοποιεί η κοινή γνώμη τόσο του Βορρά όσο και του Νότου. Πρόσφατα είχα πάει στην επισκεφτή την Φινλανδία, μια μεγάλη σημαντική πολύτιμη χώρα έχει περίπου 6 εκατομμύρια κατοίκους και όλοι αυτοί οι πολίτες έχουν ε, κοινά σύνορα με τη Ρωσία, περίπου 1.300 τόσα χιλιόμετρα. Ως εκ τούτου καλούνται να καταβάλουν στρατιωτικές προσπάθειες για να προστατεύσουν και τους ε, πολίτες ε, του νότου της Ευρώπης. Κάτι που πολλοί δεν το συνειδητοποιούν. Και το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νότος στη Μεσόγειο και ίσως θα έπρεπε να γίνει πιο συνειδητό ότι υπάρχουν κράτη που είναι εκτεθειμένα στα σύνορά μας, ε, φέρουν το βάρος της μετανάστευσης και ως εκ τούτου έχουν ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Είναι απολύτως απαραίτητο να μειωθεί η απόσταση, κυρίως απόσταση που αφορά τις Βρυξέλλες και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να λέμε ότι σε αυτή τη θητεία θα είμαστε οι επικεφαλής ε, του αγώνα της κλιματικής αλλαγής. Τι νόημα έχει αυτό εάν οι φορείς ε, των κρατών μελών δεν ευθυγραμμιστούν με την ευρωπαϊκή ατζέντα, με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Αν δεν γίνει αυτό δεν θα τα καταφέρουμε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια κοινή οπτική των πραγμάτων και επαναλαμβάνω να μειώσουμε την απόσταση γιατί σήμερα όλοι μας ε, φέρουμε μεγάλη ευθύνη. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχουμε συνειδητοποιήσει εκτός Ευρώπης ε, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στις προκλήσεις ε, που αποφάσισε να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Ως εκ τούτου, αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ε, χρειαζόμαστε όλοι να θεωρούν ότι είναι μια σημαντική ψηφίδα του μοσαϊκού, του ευρύτερου μοσαϊκού που είναι η οικονομική διακυβέρνηση ε, στην Ευρώπη, δημοκρατική οικονομική διακυβέρνηση. Αυτή λοιπόν την χρονική στιγμή αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Συγκεκριμένα υπάρχει ένα Αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητηθεί το πολιτές, ο δημοσιονομικό πλαίσιο, ο προϋπολογισμός για τα επόμενα 7 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συζητηθεί πώς θα επενδυθούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα επιτύχουμε, τι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και επίσης και πού πρέπει να γίνουν περικοπές. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση ε, θα πρέπει ε, να θεωρεί τα Εθνικά Κοινοβούλια ως ε, πρωταγωνιστές. Εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μια συγκεκριμένη οπτική για την αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δηλαδή πιστεύουμε ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα σημαντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Η γεωργική πολιτική, η πολιτική συνοχής, εάν δεν έχουμε τους απαραίτητους πόρους για να χρηματοδοτούμε τη συνοχή, τότε πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε την απόσταση ανάμεσα στα κρατη ανάμεσα στις πιο πλούσιες και τις ε, λιγότερο ευνοημένες χώρες. Την ίδια στιγμή είναι απαραίτητο να διατίθενται κονδύλια, επαρκή κονδύλια, γιατί υπάρχει αυτή η πρόκληση της Πράσινης Συμφωνίας. Και αυτό αφορά όλους. Ε, το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Αυτό είναι ένας ε, θεμελιώδης ε, στόχος γιατί οι εταιρείε μας δεν πρέπει να κλείσουν, πρέπει να μετατραπούν. Κανείς να μην χάσει τη δουλειά του, τον αντίον μάλιστα. Με την Πράσινη Συμφωνία εμείς επιθυμούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης και όχι να χαθούν θέσεις εργασίας μάχη, η συζήτηση με τα κράτη-μέλη. Βεβαίως και εσείς είσαστε πρωταγωνιστές σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς ε, δεν θέλουμε να υπάρχουν εικονικές ε, μεταφορές ε, στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, εμείς επιθυμούμε να βρούμε τη δυνατότητα έτσι ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες των κρατών μελών και ως εκ τούτου η μετάβαση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τιμωρία αλλά ως μια ευκαιρία. Αυτό, ε, αυτή είναι η πρόκληση. Αυτές τις ε, ημέρες Συζητήσαμε εκτενώς με το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το τι θα πρέπει να αποφασίσουν και να συζητήσουν οι επικεφαλείς ε, κρατών και κυβερνήσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι αν θέλουμε να μειώσουμε την απόσταση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατορθώσει, να αναπτύξει τα δικά της τα ηγετικά στελέχη, τη δική της την ηγετική θέση, για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξαναδούμε λιγάκι τους αριθμούς γιατί δυστυχώς έχουμε ανάγκη από περισσότερα κονδύλια. Και εμείς ε, θέλουμε να συζητήσουμε με εσά και να μπορούμε να ομιλούμε εκ μέρους των πολιτών. Γιατί ε, πολλές φορές ε, ο προϋπολογισμός ε, δεν γίνεται κατανοητός από τους ε, πολίτες μας. Ως εκ τούτου πρέπει να καθησυχάσουμε τους πολίτες και να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με τα κράτη-μέλη να κατορθώσει, να χαράξει μια πολιτική. Μια πολιτική έτσι ώστε να μην χαθούν θέσεις απασχόλησης, να μειωθούν οι ανισορροπίες να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταπεξέλθει ε, στις προκλήσεις που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Φέρουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή όλοι από κοινού μεγάλη ευθύνη και νομίζω ότι αυτή την ε, ευθύνη οφείλουμε να την αναλάβουμε και εδώ είναι πολύ σημαντική η δική σας η άποψη. Όσον αφορά στην κλιματική κρίση είναι μια έκτακτη ανάγκη που νομίζω όλοι το έχουν συνειδητοποιήσει. Όχι μόνο οι θεσμοί αλλά και οι πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ηγείται της παγκόσμιας δράσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κινητήρια δύναμη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ο πρώτος θεσμός που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050 και αυτό για πρώτη φορά θα ε, παγιωθεί και σε νομοθετικό επίπεδο. Αυτό θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Προφανώς και η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστική σημασίας ε, για να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας των Παρισίων και για να ε, μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να ενισχυθούν οι κλιματικοί μας στόχοι για το 2030 να μειωθούν κατά 55% οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αυτά ίσως και στην επόμενη δεκαετία. Εάν όμως θέλουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα, όπως σας είπα και προηγουμένως, όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε. Και αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή όλοι να συμμετέχουν, κανείς να μην μείνει πιο πίσω, ούτε κράτος μέλος, ούτε καμία επιχείρηση και κανένας εργαζόμενος να μην χάσει τη δουλειά του. Αυτή λοιπόν η φιλοδοξία μπορεί να σταθεί μόνο εφόσον η κοινή γνώμη στηρίξει τις απαραίτητες αλλαγές. Αλλαγές για τις κοινωνίες μας, αλλαγές για την οικονομία μας. Ως εκ τούτου οφείλουμε να εξερευνήσουμε τις ε, επιπτώσεις του προεπολογισμού, κοινωνικές επιπτώσεις ε, που θα συνοδεύουν θαραλέες πράξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πρόσφατα παρουσίασε την πρότασή της για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ιδιότητά του του συνομοθέτη καλείται να αξιολογήσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα γίνει κατά τα επόμενα δύο έτη. 50 ε, νομοθετικές προτάσεις έχουν κατατεθεί, κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα δώσουν ε, συγκεκριμένη εικόνα σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο χρειαζόμαστε τα κράτη-μέλη για να βοηθήσουν και τα κράτη-μέλη τα θεματολόγια να είναι εφικτά. Η Ευρώπη προτίθεται να αλλάξει για να ανταπεξέλθει στην πρόκληση και αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάμε την κοινωνική διάσταση των θεμάτων. Ο αγώνας κατά των ανισοτήτων ε, περιβαλλοντικές προκλήσεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο εφόσον ε, μειωθούν οι ανισότητες ε, στο κέντρο των πολιτικών μας δράσεων κλιματικές προκλήσεις και ανισότητες αυτά είναι τα προβλήματα αυτά πρέπει να έχουμε κατά νου στον αγώνα που θα δώσουμε Είμαι σίγουρος ότι οι ομιλητές μας σήμερα θα μας δώσουν ερεθίσματα για περισυλλογή. Θα κατορθώσουμε να διαμορφώσουμε ένα πολιτικό πλαίσιο για να ενταχθούν εκεί οι σκέψεις μας και για να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές θα μας επιτρέψουν να ανταπεξέλθουμε στα κλιματικά προβλήματα που καλούμεθα να επιλύσουμε. Σας εύχομαι λοιπόν ευόδοση των εργασιών σας. Ξέρω πολύ καλά ότι η συζήτηση είναι πολύ σημαντική για εσάς. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, ευόδοση λοιπόν των εργασιών και εύχομαι μαζί με μας να συνεχίσετε να είσαστε οι πρωταγωνιστές ε, όχι μόνο της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της δυνατότητας όλων των κρατών μας μελών να βρεθούν στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίω δίνω το λόγο ε, στον πρόεδρο Ράινα. Αξιότιμε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Σασόλη. Αξιότιμοι Βουλευτέ των Εθνικών Κοινοβουλίων, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Αξιότιμοι ομιλητέ, κυρία Ναβάρο, κύριε Κάρνη, κύριε Ράιντερ, κύριε Βίνκλερ, ε, κύριε Πρόεδρε της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους εγκάρδια εκ μέρους της Κορατικής ε, Βουλής και ε, εμού προσωπικά. Χαίρομαι που ε, στα πλαίσια της συζήτησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα μιλήσουμε και εδώ στην Κοινοβουλευτική Εβδομάδα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και τις συνέπειές τους στις οικονομικές, κοινωνικές και δημοσιονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι συμφωνούμε στο ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και ακριβώς η δική μας η γενιά θα πρέπει να υπομειστεί αυτή την ειδική ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το 10% των παγκόσμιων ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα έχει τη φιλοδοξία να γίνει παγκόσμιο ηγέτη τη καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών με τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τι επενδύσει στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και την υλοποίηση τη κλιματική ιδιωτερότητα μέχρι το 2050, όπω ανέφερε και ο πρόεδρο όλοι πριν από λίγο. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα εγγενιάσουμε ένα νέο κύκλο ρηξικέλευθων αλλαγών και αυτό το σχέδιο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως σχέδιο μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η οικολογική μετάβαση έχει τεράστιο δυναμικό για την οικονομική ανάπτυξη με νέα επιχειρηματικά μοντέλα αγοράς, περισσότερες θέσεις απασχόλησης, τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και όλα αυτά προσανατολισμένα προς το μέλλον. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα κράτη-μέλη που δεν έχουν το ίδιο σημείο αφετηρίας ε, θα είναι δύσκολο να περάσουν σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ε, σημαντική αλλά δίκαιη και ισορροπημένη μετάβαση ώστε όλοι να απολαύσουν ισότιμους κανόνες και ισότιμες συνθήκες. Και γι' αυτό θα μας χρειαστεί ε, τεράστιος βαθμός και δημόσιων αλλά και ιδιωτικών επενδύσεων. Και αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στις τρέχουσε διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπει ε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Έναν μηχανισμό για τη δίκαιη μετάβαση θα έπρεπε να κινητοποιήσουμε περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ για τις περιφέρειες και τους πολίτες που θα πληγούν περισσότερο από τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει συστημικές αλλαγές και αλλαγή και της νοοτροπίας, του τρόπου σκέψης αλλά και του τρόπου διαβίωσης μερικές φορές, του στυλ ζωής μας. Και ε, αυτό θα ε, απαιτήσει τεράστιες δεσμεύσεις και προσπάθειες από όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κροατία ως χώρα με πολύ φυσικό πλούτο αναγνωρίζει τη σημασία αυτού του φιλόδοξου σχεδίου της Νέας Πράσινης Συμφωνίας και εστερνιζόμαστε τους, σκόπους, τους στόχους αυτούς με τη στρατηγική μας για την ενέργεια μέχρι το 2030 ενώπιση της πολιτικής για το 2050 και ε, με τα ολοκληρωμένα σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030. Εμείς ε, τονίσαμε την ε, ανάγκη εξασφάλισης του ενεργειακού ανεφοδιασμού αλλά και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις εκπομπές των καυσερίων, των αερίων του θερμοκηπίου και μέχρι στιγμής βρισκόμαστε πάνω από το κοινότικό μέσο σε ό,τι αφορά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών πηγών ενέργειας και την, ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ανακάτοικο. Ε, η Κροατία το 38% των ενεργειακών της αναγκών ε, τις ικανοποιεί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περίπου περάσαμε από το 20% στο 40% και μάλιστα βρισκόμαστε στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή την άποψη. Βέβαια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποιε οικονομικέ συνέπειε και αυτό που προβληματίζει κυρίω του συμπολίτε μα, που είναι οι δαπάνε. Σίγουρα θα χρειαστούν ε, περισσότερε δαπάνε και επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγέ ενέργεια. Γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερο πρόγραμμα στήριξη ε, των νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή ένδια για να βελτιωθεί το βιωτικό του επίπεδο. Θα θα πρέπει λοιπόν να του αφήσουμε πίσω. Σα ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε μου τώρα να καλωσορίσω καλωσορίσω τον πρώτο μας ομιλητή, τον κύριο Μάρκ Κάρνι που είναι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την πολιτική για το κλίμα και τη χρηματοδότηση. Κύριε Κάρνι, παρακαλώ έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Θα μιλήσω κυρίως για το πόσο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να ενισχύσει ...της δράσης του δημοσίου τομέα για το κλίμα. Αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσω τη σημασία της κρίσης, της μεγάλης προσδοκία και να πω ότι φέτος πρέπει να αναλάβουμε δράση. Η COP26 που θα φιλοξενήσουν η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια κρίσιμη ευκαιρία να βάλουμε τις εκπομπές σε μια πορεία περιορισμού. Σύμφωνα με την COP25, όπως ξέρει και το Κοινοβούλιο, αυτό ένα ουδέτερο ισοζύγιο, η μετάβαση δηλαδή, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία του καιρού μας. Ο στόχος της COP26 είναι πολύ απλός. Κάθε οικονομική, κάθε χρηματοπιστωτική απόφαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κλίμα. Αυτό αφορά τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τις ε, πολυμερεί αναπτυξιακές τράπεζες και ιδίω τον ιδρυτικό τομέα. Η στρατηγική μας για την COP26 ξεκινά με μια απλή πρόταση. Δεδομένου ότι το ουδέτερο ισοζύγιο είναι το ελάχιστο, ελάχιστος κοινό ε, παρομαστής, πρέπει να δείξουμε τον δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλοι είναι η υπέρτατη ανάγκη που προκύπτει από την φυσική ανάλυση του κλίματος. Κάθε εταιρεία, κάθε επιχείρηση, κάθε συνταξιδοτικό ταμείο, κάθε ιδρυτικός φορέας, κάθε κυβέρνηση πρέπει να καταστρώσουν σχέδια για ουδέτερο ισοζυγείο. Και για να δούμε ποιος είναι έτοιμος και ποιος όχι, και για να διαπιστώσουμε πού βρίσκονται οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες, πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο σε τρει τομεί. Αναφορά, διαχείριση κινδύνου και απόδοση. Από όλε όμω τι απόψει, ο ηγετικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμβολή αυτού του Κοινοβουλίου θα διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο. Και ξεκινώ με την ε, δημοσιοποίηση. Ένα παλιό αξίωμα λέει ότι μόνο αυτό που μπορεί να μετρηθεί μπορεί να τύχει διαχείριση. Στο Παρίσι πριν από χρόνια οι ηγέτε του G20 δημιούργησαν την TCFD που αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που επηρεάζουν το κλίμα. 18 μήνες αργότερα, στο Αμβούργο, στο G20, η Επιτροπή αυτή υπέβαλε συστάσεις για τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν το κλίμα. Σήμερα, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείε, ε, ταμεία, επενδυτές κλπ. που εκπροσωπούν 135 εκατομμύρια, το παραλαμβάνω, 135 εκατομμύρια δολάρια, ζητούν τέτοιου είδου στοιχεία από τις επιχειρήσεις. Στην COP26 στη Γλασκόβη σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια συμμαχία αρχών, οργανισμών που ενδιαφέρονται για το κλίμα και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και θα καταστήσουν την πρακτική αυτή υποχρεωτική. Και θέλουμε βεβαίω οι δεσμεύσει αυτέ να είναι δεσμευτικές και ολοκληρωμένε κατά το δυνατόν. Θα ήθελα με την ευκαιρία να συγχαρώ και πάλι την ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν υιοθέτησε τι σχετικέ κατευθυντήριε γραμμέ πέρσι σχετικά με τη δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων και ο αντιπρόεδρο των Πρόφσκη ε, προχθέ αναφέρθηκε στι δημοσιοποιήσει αυτέ ω ακρογωνιαίο λίθο των υποχρεώσεων δημοσιοποίηση χρηματοπιστωτικών στοιχείων που επηρεάζουν το κλίμα και ότι θα ενσωματωθούν αυτά στη σχετική οδηγία. Καθώς λοιπόν θα αναπτύσσονται όλα αυτά και η σχετική οδηγία περί δημοσιοποίησης στοιχείων, να ξέρετε ότι και η TCFD συνεχίζει να προοδεύει προς τα εμπρός και να ξέρετε ότι πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο πρότυπο δημοσιοποίησης στοιχείων όσον αφορά το κλίμα και αφορά την διαχείριση του κλίμα, τη διαχείριση του κινδύνου με τρόπο μετρήσιμο. Συμμετέχει ο ιδρυτικός τομέας, και συγκεράζονται εκεί οι απόψεις των επιχειρήσεων που ζητούν χρηματοδότηση αλλά και αυτών που χορηγούν κεφάλαια σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η συμμαχία αυτή υποστηρίζεται από τις συστημικές τράπεζες και από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 90% των διχειριστών περιουσιακών στοιχείων, από συμβούλους, επενδυτών και ούτω καθεξής. Το αντικείμενο είναι λοιπόν η υπεύθυνη επένδυση. Όλοι συμφωνούν ότι η αυτή πρέπει να γίνει το πρότυπο το οποίο θα επικρατήσει. Θα συνεργαστούμε μαζί σας καθώς προχωρούμε προς τα εμπρός με σκοπό ένα ενιαίο πρότυπο δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν το κλίμα. Και τώρα, όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου, ο δρόμο για την εφορική χρηματοδότηση περιλαμβάνει βεβαίω και την διαχείριση κινδύνου και αυτό απαιτεί δημοσιοποίηση στοιχείων ε, όχι στατικών, όχι αυτά που δημοσιεύουν σήμερα οι επιχειρήσει σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα. Χρειαζόμαστε σχέδια για την μείωση αυτών των εκπομπών. Διαχείριση κινδύνου σημαίνει να αξιοποιήσουμε, να αξιολογήσουμε μάλλον τα σχέδια που έχουν επιχειρήσει καταστρωμένα για τη μείωση του αποτυπώματο. Και αυτό σημαίνει τεστ αντοχή. Η Τράπεζα τη Αγγλία μάλιστα πέρσι έγινε η πρώτη κεντρική τράπεζα η οποία υποδεικνύει λύσεις στους τέρους της για μια ομαλή μετάβαση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να πετύχουμε όλοι. Στόχος είναι λοιπόν ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, χωρίς μερικές δεν θέλουμε να φτάσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα καταστροφικό σενάριο. Οι δοκιμέ λοιπόν αντοχή στι τράπεζε, αλλά και στι επιχειρήσει που ετοιμάζονται για την μετάβαση προ το δεύτερο ισοζύγιο θα εκθέσουν αυτού οι οποίοι ακόμη δεν έχουν καταστρώσει μια σχετική στρατηγική. Η Τράπεζα της Αγγλίας θα συνεργαστεί με άλλες, ήδη μάλιστα συνεργάζεται με άλλες 50 κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές ανά τον κόσμο ώστε η τεχνολογία αυτών των ε, δοκιμών αντοχής να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερομένους και εδώ για άλλη μια φορά χαιρετίζουμε τον ηγετικό ρόλο της ESRB και της EAB και άλλων συστημικών τραπεζών στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που υποστηρίζουν αυτές τις δοκιμές αντοχής. Να προσθέσω επίσης ότι αυτές οι δοκιμές αντοχής όχι μόνο αποκαλύπτουν πώς διαχειρίζονται οι τράπεζε του κινδύνου, αλλά και πώ τονώνεται η ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού μα συστήματο και γίνονται πιο αποδοτικέ οι πολιτικέ για το κλίμα. Τρίτο θέμα, τρίτο πυλώνα, η απόδοση, οι αποδόσει. Έλεγα ότι η μετάβαση σε ουδετερό ισοζύγιο είναι μια τεράστια οικονομική ευκαιρία. Είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει, θα έχει αντίκτυπο σε κάθε, σε κάθε τομέα οικονομική δραστηριότητα. Και δεν είναι μόνο να υποστηρίξουμε τι πράσινε τεχνολογίε. Καλό αυτό. Όμω, οι εταιρείε οι οποίε είναι στη μετάβαση πρέπει να επιβραβευθούν. Γιατί ο κόσμος ζητά δράση για το κλίμα. Πρέπει λοιπόν τα ταμεία, οι ασφαλιστικέ πρέπει να αποκαλύψουν σήμερα, να δημοσιοποιήσουν πώ αξιοποιούν τα χρήματα των πολιτών, των συνταξιούχων, των επενδυτών και ότι το κάνουν σύμφωνα με τις αξίες τους. Η απλή λοιπόν καταγραφή δεν είναι επαρκής. Καλή δράση λοιπόν για το κλίμα, τη διακυβέρνηση, την κοινωνία. Τι γίνεται συγκεκριμένα όμω με τη μεταβολή του κλίματο και τι σκοπεύετε να κάνετε. Το να καταγράφουμε απλώ τι εκπομπέ μα δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Και η κατηγοριοποίηση βεβαίω των εκπομπών είναι και αυτή ένα καλό βήμα, όμω σα προειδοποιώ ότι μπορεί να φτάσουμε να δημιουργήσουμε μια μαύρη λίστα ε, επιχειρήσεων, χωρίς όμως να έχουμε επιτύχουμε τη μετάβαση και χωρίς να επιβραβεύουμε αυτούς που κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι οι επενδυτέ, οι των κεφαλαίων να προετοιμαστούν και αυτοί για την λεγόμενη μετάβαση προς το ουδέτερο ισοζύγιο. Το πιο βασικό μέγεθος είναι τι ποσοστό των κεφαλαίων επενδύεται σύμφωνα με τις αρχές της TCFD. Ένα άλλο βήμα θα ήταν να αξιολογήσουμε το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που συνάδουν με τις αρχές των Παρισίων. σε ποιε επιχειρήσει δηλαδή επενδύεται και είναι αυτέ σε περίοδο μετάβαση. Και τέλος, έχουμε τον στόχο βεβαίω ε, για την κατηγορία 3 εκπομπών. Ζητάμε επίση ε, λεπτομέρειε όσον αφορά την διακυβέρνηση, εάν οι αμοιβέ των στελεχών ε, συναρτώνται με τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έχουν σχέση με το κλίμα. Και εν τέλει έχουμε τον συγκερασμό αυτών των πληροφοριών για να αξιολογήσουμε το κατά πόσον και σε, κατά πόσους βαθμούς Κελσίου η δράση της χ επιχείρησης συμβάλλει στην θέρμανση του πλανήτη. Η Διαξά, η Αλιάνς δημοσιοποιούν εθελοντικά αυτές τις πληροφορίες στην πορεία προς την COP26. Ω την COP26, ο σκοπό είναι οι επιτυχίε αυτών των προσεγγίσεων να αξιοποιηθούν και να έχουν διαμορφώσει μια συμμαχία ιδιοκτητών περιουσιακών στοιχείων, επενδυτών και επιχειρήσεων που δανείζονται για να φτάσουμε όλοι μαζί στο ουδέτερο ισοζύγιο. Και εδώ θα χρειαστούμε τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να εφαρμόσουμε αυτήν την προσέγγιση στις πολυμερείς ε, επενδυτικέ τράπεζε. Να μην έχετε λοιπόν καμία αμφιβολία. Οι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πετυχαίνουν ήδη. Ο συνδυασμό τη κρίση του κλίματο, τα αιτήματα του κοινού, ο στόχος του ουδετερού ισοζυγίου. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι προσδοκίες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλάζουν και αυτές. Και όπως έλεγε και κάποιος πρόσφατα, η αηφορική χρηματοπιστωτική δραστηριότητα είναι το νέο ίντερνετ, επηρεάζει κάθε επιχείρηση και κάθε επενδυτικό κεφάλαιο. Ας αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία. Το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι στα πρώτα απέχουμε πολύ όμω από το να υλοποιήσουμε την υπόσχεσή μα. Οι εθελοντικέ δράσει που παρατηρούμε είναι καλοδεχούμενε βεβαίω, αλλά χρειάζεται περαιτέρω συντονισμό από τι κυβερνήσει και από τα κοινοβούλια. Ο δημόσιο τομέα έχει μια ευκαιρία να καθοδηγήσει τον ιδιωτικό τομέα. Και η ευκαιρία δεν θα είναι εδώ για πάντα. Η εφορική χρηματοπιστωτική ε, δράση ξεκινάει μόλις τώρα, όμως έχουμε ήδη καθυστερήσει ο πλανήτης υπερθερμαίνεται, οι υπολογισμοί έχουν γίνει συνολικά για τον πλανήτη, πλανήτη με συγχωρείτε, περιμένουμε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη περίπου 3,5 βαθμού σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Και έχουμε και την πίεση της κοινή γνώμης. Η κοινή γνώμη βρίσκεται μπροστά από αυτά τα οποία κάνουν οι κυβερνήσει. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμένη δράση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Γιατί η κοινή γνώμη, όπω είπα, πιέζει ε, και δεν θέλουμε να φτάσουμε σε υπεραπλουστικές λύσεις όπως η αποεπένδυση ή άλλες ρητικές λύσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Εν κατακλείδη λοιπόν χρειάζεται δράση. Η δράση αυτού του κοινοβουλίου θα βοηθήσει, θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο και ας αξιοποιήσουμε την COP26 και την Προεδρία της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για να τονώσουμε τις προσπαθειές μας και να διαμορφώσουμε εκείνες τις μαχίες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να δράξουμε τις ευκαιρίες και να κάνουμε κάτι επιτέλους για το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ. Um, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα είμαι εγώ η συντονίστρια στις υπόλοιπες συζητήσεις που ελπίζω να είναι ζωηρές. Ε, όπως ε, είπε ο κύριος ε, Μακάρνη, έχουμε 50 αποχρώσεις του πρασίνου. Εμείς είχαμε 40 στην Ιρλανδία, οπότε ήδη υπάρχει αύξηση των αποχρώσεων. Θα δώσω το λόγο στον Γκάι Ράιντερ, το Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, για μια δεκάλεπτη παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας το, το Κοινοβούλιο και την Κροατική Προεδρία που μα έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω σήμερα. Ε, ο Διεθνής Οργανισμός ε, Εργασίας ε, έχει εμπνευστεί από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεργασία αυτή ήταν επιτυχημένη μόνο γιατί βασιζόταν σε κοινέ αξίες, στην κοινωνική δικαιοσύνη, σε κοινέ μεθόδους, στις κοινωνικές συνεργασίες στον διάλογο και διότι όλοι ήμασταν πρόθυμοι να αγκαλιάσουμε νέε προκλήσει και ευκαιρίε. Σήμερα ε, η ΑΕΛΟ, Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασία ε, προχωράει μετά την εκατονταετηρίδα και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινούν ένα πολύ ε, φιλόδοξο πρόγραμμα. Καλούμεθα λοιπόν να συνεργαστούμε να επιτύχουμε ένα καλύτερο, περισσότερο βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη και τον κόσμο. Για είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι τον Οκτώβρη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσόρισε την διακήρυξή μας για το μέλλον της εργασίας. Αυτή υιοθετήθηκε τον Ιούνιο και ε, αναφέρεται με μεγάλη ικανοποίηση ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι ε, ανθρωποκεντρική. Η διακήρυξη ε, προσφέρει ένα νέο χάρτη, μια νέα πορεία στις εσωτερικές και τις εξωτερικές πολιτικές. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω θερμά τη δέσμευση για την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι εξακολουθούν να αμφισβητούν το ότι η κλιματική αλλαγή είναι το αποτέλεσμα τη ανθρώπινη δραστηριότητα. Όμω πολλοί ξεχνάνε ότι σε μεγάλο βαθμό η ε, δραστηριότητα αυτή ε, βασίζεται στη δική μα δουλειά, άρα είναι και δική μα υπόθεση. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει. Ε, ο Γενικό Γραμματέα των ΗΕ σε κάθε ευκαιρία μα υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή προχωράει πολύ πιο γρήγορα από τι προσπάθειε μα να την αναχαιτήσουμε κλείσουμε Η COP25 στη Μαδρίτη ε, απλά σημαίνει ότι έχουμε καθυστερήσει ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε ήδη τις συνέπειες. Από το 2000, ε, μεταξύ 2000 και 2015 χάθηκαν περίπου 23 εκατομμύρια χρόνια εργασίας ε, ανθρώπινης ζωής και αν στρέψουμε το βλέπω στο μέλλον θα δούμε ότι οι δικές μας οι προβλέψεις μέχρι το 2030 ε, θα σημαίνουν αν συνεχίσουμε με δύο τρόπο το 2% ορών εργασία θα μπορούσαν να χαθούν γιατί απλά θα είναι πάρα πολύ ζεστό το κλίμα για να δουλέψει κανεί σε κάποιε χώρε. Μιλάμε δηλαδή για 72 εκατομμύρια θέσεις απασχόληση, πλήρου απασχόληση. Βρισκόμαστε λοιπόν σε σημείο καμπή ε, και φοβούμαστε ότι θα έχουμε ανεπανόρθωτέ ζημιέ. Ε, το ίδιο, σημείο, το ίδιο ισχύει και για την κοινή γνώμη. Πρόσφατα ε, πολλοί που συνθέτουν την ΑΕΛΟ, οι κυβερνήσει, οι εργοδότε, οι εργαζόμενοι είπαν ότι αν καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα στις θέσεις απασχόλησης και την ανάπτυξη ε, και την βιώσιμη ε, ανάπτυξη από την άλλη, τα νέα είναι πολύ καλά γιατί ε, όχι μόνο έχει γίνει κατανοητό ότι δεν μπορούν να υπάρχουν θέσει απασχόλησης σε ένα νεκρό πλανήτη, αλλά και επίση και η μετάβαση στην ε, ουδετερότητα, κλιματική ουδετερότητα γίνεται όλο και πιο απαραίτητη. Εμείς πιστεύουμε ότι 18 εκατομμύρια θέσει απασχόληση μέχρι το 2030, 24 εκατομμύρια έχουν ήδη συσταθεί και 6 εκατομμύρια έχουν χαθεί. Αυτά είναι ο στόχο εάν κάνουμε το σωστό στην Ευρώπη που είναι ε, να μειώσουμε ε, κατά 2% τη θερμοκρασία, αυτό που αναφέρεται στη Συμφωνία των Παρισίων. Και έτσι θα προκύψουν πολλέ θέσει. Απασχόληση κυρίω στον τομέα των κατασκευών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Εναλλακτικό λοιπόν σενάριο στην αποκάλυψη, ε, αυτό θέλουμε όλοι μα, αλλά δεν θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε απλά ε, διακηρύσσοντάς το. Ε, χρειαζόμαστε και μια ουσιαστική πολιτική και ακριβώ εδώ έρχεται η Πράσινη Συμφωνία. Θέλω γρήγορα να υπογραμμίσω δύο στοιχεία τη πράσινη συμφωνία που κατά την άποψή μου είναι καθοριστική σημασία. Πρώτον, η Ευρώπη δεσμεύεται για μια δίκαιη μετάβαση. Ο πρόεδρος κύριος Σασόλη υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι όλοι ίσοι ε, όσον αφορά την οικολογική κρίση και ότι οι προκλήσεις ε, του κλίματος και της ανισότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο αν είμαστε ενωμένοι. Γι' αυτό λοιπόν η στρατηγική της Ευρώπης βάζει τον άνθρωπο στην πρώτη θέση με προτεραιότητα στις περιφέρειες, στις βιομηχανίες, στους εργαζόμενους που θα αντιμετωπίσουν τα περισσότερα προβλήματα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πιστεύω ότι αν δεν είναι δίκαιη η κλιματική μετάβαση απλά δεν θα λάβει χώρα γιατί θα είναι αντίθετη με την λαϊκή άποψη και οι πολίτες θα τη σταματήσουν και θα δούμε γεγονότα στην Ευρώπη είδαμε και κάποια πρόσφατα που στηρίζουν αυτό που λέω βεβαίως εύκολα μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι παράλογα είναι αυτοκτονικά αλλά είναι πραγματικά εκπλήσει το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι των οποίων ε, το βασικό που του απασχολεί στη ζωή του είναι να φτάσουν μέχρι το τέλο του μήνα, να μπορούν να επιβιώσουν. Ε, Θεωρείτε ότι είναι ε, υπερβολικό το να ανησυχούν αυτοί για το τέλο του πλανήτη. Οι πολίτε πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα βρεθούν μόνοι του μπροστά σε αυτό το δίλημα. Το μήνυμα έχει ακουστεί, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίε. Το Σεπτέμβρη είχαμε συνάντηση κορυφή στα Ηνωμένα Έθνη και ο γενικό Γραμματέας ξεκίνησε μια πρωτοβουλία, η ΑΕΛΟ ανέλαβε πρωτοπόρο θέση και 46 χώρες έχουν ήδη υπογράψει για μια δίκαιη μετάβαση αυτή να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των βιώσιμων προγραμμάτων ανάπτυξης. Ως εκ τούτου αυτό που κάνει η Ευρώπη με την Πράσινη Συμφωνία το κάνει και ο υπόλοιπο κόσμος. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του θεματολογίου 2030 βιώσιμη ανάπτυξη και η Ευρώπη έχει δεσμευτεί σε αυτό το θεματολόγιο. Εάν λοιπόν ο πρωταρχικός στόχος είναι όλοι να συμμετέχουν στη μετάβαση για την κλιματική ουδετερότητα, κανείς δεν πρέπει να εξαιρείται στο σχεδιασμό του δρόμου προς τα εμπρός. Εδώ η Ευρώπη έχει θαυμάσια εργαλεία ε, στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, κυρίως αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων που είναι και ε, εταίροι σε οτιδήποτε κάνει η ILO. Το δεύτερο, η Πράσινη Συμφωνία αναγνωρίζει ότι η κλιματική μετάβαση απαιτεί μεγάλες επενδύσεις ε, και έχει διατάξεις για, τις, για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Και όλα αυτά γίνονται μέσα από ένα συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και με το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Εσείς λοιπόν ε, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αποφασίσετε κατά πόσον ε, τα κονδύλια που προτείνονται είναι επαρκή. Αλλά και εδώ είναι απαραίτητο η παγκόσμια δράση να αντικατοπτρίζει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Ο Μαρκ Κάρνι έχει γίνει ειδικό απεσταλμένος των ΗΕ για την κλιματική δράση και τα χρηματοοικονομικά και αυτό είναι μια πολύ καλή εγγύηση. Ακούσατε ε, την μαρτυρία του προηγουμένως. Ε, εγώ θέλω απλά να προσθέσω κάτι σε αυτά που ήδη μας είπε. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και στις δικές μας συζητήσεις για την εργασία και το κλίμα. Πρόκειται απλά για το ότι αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες οι οποίες αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα ε, της συμμετοχής μας στην Ευρώπη και αλλού έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ευημερίας μόνο επειδή μπορεί και ακολούθησαν ένα αρνητικό δρόμο που τώρα στρέφεται εναντίον τους. Νομίζω λοιπόν πρέπει να γίνει αυτό κατανοητό. Όχι μόνο διότι πλήττονται, περισσότερο οι αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και διότι ε, αυτό δείχνει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πια ε, να ξεχάσει ε, το τι συνέβη και να προχωρήσει προς τα εμπρός, θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικέ λύσεις. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Πρόεδρε, η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις εξωτερικές αλλά και εσωτερικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα δεν μπορούμε να κερδίσουμε από μια Ευρώπη ουδέτερη σε άνθρακα εάν στον κόσμο εξακολουθεί να γίνεται χρήση των ορυκτών καψίμων. Ε, η Πράσινη Συμφωνία μπορεί λοιπόν να κάνει κάτι το οποίο ε, μέχρι τώρα δεν ήταν εφικτό. Και τι είναι αυτό, είναι να περάσει το τεστ της αξιοπιστίας. Να πιστούν οι άνθρωποι ότι θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον σε ένα κλιματικά ουδέτερο κόσμο. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω έτσι χαρακτηριστικά γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά. Το 2008 στο περιθώριο της COP14 στην Πολωνία συναντήθηκα με συνδικαλιστές σε ορυχείου στη Σιλεσία και τους μίλησα για την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, στην πάψη χρήση των ορυκτών καυσίμων και μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν τους έπεισα και είμαι σίγουρος ότι ούτε και εγώ πίστηκα. Γιατί, διότι τότε δεν υπήρχε αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Ε, τι δίκαιη μετάβαση, δεν υπήρχαν επενδύσεις, δεν υπήρχε μέλλον για αυτούς. Αυτό λοιπόν είναι το κλασικό λάθος που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επαναληφθεί. Χρειαζόμαστε αξιόπιστη μετάβαση για ένα καλύτερο μέλλον. Η διακήρυξη εκατονταετίας ε, της ILO για το μέλλον της εργασίας ε, ε, που εγκρίθηκε όπως σας είπα τον Ιούνιο προβλέπει ένα μέλλον ε, με διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης και είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας ε, θα βασιστούν ε, σε αυτή την μακροχρόνια συνεργασία που είχαν μέχρι σήμερα. Πολύ σημαντικό για να αντιμετωπιστεί το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Ράιντερ. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω την τρίτη μας ομιλήτρια, την κυρία Έλενα Ναβάρο, που είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και να της δώσω το λόγο για ένα δεκάλεπτο επίσης. Παρακαλώ κυρία Ναβάρο. Καλημέρα σας. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση και να αναγνωρίσω τον κέριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων στη μετάβαση που επιχειρούμε προκειμένου να καταστήσουμε την Ευρώπη την ε, πρώτη ε, ήπειρο στον κόσμο με ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα. Είναι σαφής ο προορισμός μας. Ε, κλιματική ουδετερότητα με δίκαιη μετάβαση που δεν θα αφήνει κανέναν ουραγό, κανέναν αποκλεισμένο. Και αυτό είναι σημαντικό για του πολίτε, ιδιαίτερα για την ε, γενιά. Και αυτή είναι η απέτηση των πολιτών. Κατεπίγουσε δράσει για να ανταποκριθούμε στην έκτακτη ανάγκη για το κλίμα. Ετοιμάζουμε τώρα τον οδικό χάρτη για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και πολύ σύντομα θα έχουμε την Ευρωπαϊκή ε, Νομοθεσία για το κλίμα για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και να μην αποκλίνουμε από την πορεία μας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι και είναι ε, σαφές ε, ότι η πορεία μας ε, θα είναι γεμάτη δύσκολες επιλογές και προκλήσεις. Η απαλλαγή από τον άνθρακα της οικονομίας μας είναι μια περίπλοκη διαδικασία που θα απαιτήσει ριζικό μετασχηματισμό των οικονομιών και των τρόπων ζωής μας. Όπως μας υπενθύμησε ο κύριος Κάρνη, τα χρηματοοικονομικά και η χρηματοδότηση θα παίξουν ένα θεμελιώδη ρόλο για την υλοποίηση της μετάβασης και αυτός είναι και αυτό είναι το περιεχόμενο της ομιλίας μου. Ο ρόλος της χρηματοδότησης και το έργο της ΕΤΕΠ προκειμένου να στηρίξει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες και να αποτελέσει βασικό εταίρο στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Είναι τεράστιο το κενό που έχουμε στι χρηματοδοτήσει στι περιβαλλοντικέ. Χρειαζόμαστε τεράστιε επενδύσει για να απαλλαγούμε από τον άθρακα στι οικονομίε μα και να αναπτύξουμε νέε τεχνολογίε που θα έχουν ε, κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση και στη διευκόλυνση αυτή τη μετάβαση και του μετασχηματισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε ότι για να υλοποιήσουμε του στόχου για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 θα, θα απαιτήσει 260 επιπλέον ε, δισεκατομμύρια το χρόνο πλέον επιπλέον επενδύσεις και ε, αυτό δεν λαμβάνει καν υπόψη τα σχέδιά μας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και για την αύξηση των αρχικών ε, στόχων μας ε, και των γενικότερων κλιματικών μας και περιβαλλοντικών μας στόχων. Κανένα κράτος από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες. Οι εταιρείε και τα νοικοκυριά θα πρέπει φυσικά να χρησιμοποιήσουν το σύνολο αυτών των κεφαλαϊκών δαπανών. Αλλά χρειαζόμαστε γι' αυτό ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα κατευθύνει τι ε, ε, κεφαλαϊκέ ροέ προ βιώσιμα προγράμματα. Ένα σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη και κλιματικά κριτήρια και θα καθοδηγήσει τους επενδυτές προς τα σωστά και βιώσιμα σχέδια. Εν ολίγης, θα πρέπει να θέσουμε τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των επενδυτικών μας αποφάσεων. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται με διάφορες ε, πρωτοβουλίες στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για τη βιωσιμότητα δίνοντας στους επενδυτές περισσότερες πληροφορίες και βοηθώντας τους να κάνουν εμπεριστατωμένε αποφάσεις για βιώσιμες επενδύσεις. Με την πρωτοβουλία αυτή θα αναπτύξουμε αξιόπιστα στοιχεία και θα θέσουμε κοινά πρότυπα και προδιαγραφές που είναι απαραίτητα όχι μόνο για να προωθήσουμε τις φιλοπεριβαλλοντικέ επενδύσει, αλλά και για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό στην Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών. Η ταξινομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των πράσινων επενδύσεων για να αποφύγουμε το πράσινο ξέπλυμα στις αγορές. Πώς θα στηρίξουμε όμως αυτό το εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης σε τεχνικό επίπεδο. Ε, χαιρετίζουμε την πολιτική συμφωνία του Δεκεμβρίου των ε, συνομοθετών και ήδη ε, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε την ταξινομία και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε συμβουλές για την ανάπτυξη καταξιδότηση πράξεων στα πλαίσια της νέας πλατφόρμας για, τις, για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά. Πέραν όμως του νομοθετικού πλαισίου, ήδη διαπιστώνουμε κάποια, κάποιες ελπιδοφόρες αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Και μάλιστα οι διαχειριστές κονδυλίων ήδη συμπεριλαμβάνουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια κυβέρνησης στις επενδυτικές του στρατηγικές. Και κάποιες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ήδη έχουν αρχίσει και επενδυτικές επιχειρήσεις να ε, μειώνουν τα περιουσιακά της στοιχεία που στηρίζονται στον άνθρακα. Και οι κεντρικές τράπεζες και οι επόπτες Επίσης, ε, ε, λαμβάνουν υπόψη το κίνδυνο σε σχέση με το κλίμα στις δράσεις τους και ετοιμάζουν κλιματικά τεστ αντοχής. Το κλίμα θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην επερχόμενη ε, αναθεώρηση της ε, νομισματικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένω ακροάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ε, πρόεδρος Λαγκάρτ. Και ιδιωτικέ αλλά και πολυμερει τράπεζε, θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην άντληση κεφαλαίων που χρειάζονται για να χρηματοδοτηθεί η μετάβαση. Και έτσι μπορούμε να έχουμε βιώσιμες επενδύσεις που έχουν αποδείξει το δυναμικό τους, την ευκαιρία τους και, την, και τα ε, ωφέλη τους. Έτσι θα αξιοποιήσουμε τον καταλητικό ρόλο που μπορεί να δημιουργήσει η ΕΤΕΠ. Και τέτοιες βιώσιμες ε, επενδύσεις μπορούν να καταστήσουν κάποια πιο επικίνδυνα ε, από άποψη κινδύνου σχέδια πιο ελκυστικά και πιο αποδοτικά για να προσελκύσουν και οι ιδιώτες επενδυτές. Στην περίπτωση της ΕΤΕΠ η πορεία μας είναι σαφής και έχουμε δεσμευθεί στεναρά να συμβάλλουμε όσο μπορούμε για να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να χρηματοδοτήσουμε τη μετάβαση προς ένα θεκτικό μέλλον με χαμηλό άνθρακα. Είμαστε η τράπεζά σας, η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα χρειαστούν σημαντικές επενδύσεις για την ευημερία, τη μελλοντική μας ασφάλεια και ευημερία και είμαστε έτοιμοι να τη στηρίξουμε και δεν ξεκινούμε εκ του μηδενό. Η κλιματική δράση εδώ και καιρό αποτέλεσε ύψη προτεραιότητα των δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ ε, παράλληλα με την ευρωπαϊκή ηγεσία στο θέμα αυτό. Και από το 2012 έχουμε παράσχει πάνω από 170 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης για κλιματικές δράσεις και περιβαλλοντικά σχέδια παγκοσμίω. Επιπλέον έχουμε στηρίξει πάνω από 600 δισεκατομμύρια επενδύσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Ε, ε, έτσι έχουμε γίνει από τους μεγαλύτερους παγκοσμίους πολυμερείς παρόχους και χρηματοδότες ε, ε, κλιματικής δράσης. Επίσης είμαστε οι πρώτοι που έχουμε ε, εκδώσει κλιματικό ομόλογο το 2007 και έχουμε αναπτύξει αυτή την αγορά των πράσινων ομολόγων που έχει μεγάλο δυναμικό. Και παρά το ιστορικό μας υπέρ της κλιματικής αλλαγής, είναι σαφές ότι η κλίμακα των σημερινών προκλήσεων απαιτεί πολύ μεγαλύτερε φιλοδοξίε. Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό και πέρυσι τον Νοέμβριο αποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε τι κλιματικέ μα δεσμεύσει και φιλοδοξίε και να διατρανώσουμε το ρόλο μα ω η κλιματική τράπεζα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι μα στόχοι είναι σαφεί. Καταρχήν, δεσμευτήκαμε να αυξήσουμε το μερίδιο τη κλιματική και περιβαλλοντική χρηματοδότηση στο 50% των δραστηριοτήτων μα μέχρι το 2025. Έτσι θα ε, προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ επενδύσεων για τους στόχους αυτούς παγκοσμίω την επόμενη δεκαετία που θα είναι και η πιο κρίσιμη. Αυτός ο στόχος είναι εφικτός, αν και αρκετά δύσκολος. Πέρυσι χρηματοδοτήσαμε πάνω από 21 δισεκατομμύρια ευρώ κλιματικών και περιβαλλοντικών σχεδίων. Το 34 δηλαδή τα 100 του συνολικού δανεισμού της ΕΤΕΠ. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό σημείο αφετηρίας. Η δεύτερη μας δέσμευση είναι να ευθυγραμμίσουμε όλες τις χρηματοδοτικές μας δραστηριότητες με τις αρχές και στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων μέχρι τα τέλη του 2020. Η δέσμευση αυτή είναι πολύ σημαντική. Γιατί δεν έχει νόημα να, από τη μια να έχουμε σημαντικό κλιματικό έργο και από την άλλη να υπονομεύουμε και να υποσκάπτουμε τις προσπάθειές μας. Γι' αυτό αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε ενεργειακά σχέδια, να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε ε, ενεργειακά σχέδια που στηρίζονται σε ορυκτά καύσιμα και φυσικό αέριο μέχρι το τέλ, τα τέλη του 2021. Και είμαστε η πρώτη πολυμερής τράπεζα που υιοθέτησε τέτοια απόφαση. Ένα άλλο κρίσιμο σημείο της νέας κλιματικής στρατηγικής μας είναι η υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης και σε τελική ανάλυση, η κλιματική δράση και η η μετάβαση θα πρέπει να θεωρηθούν ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αναφέρθηκε και ε, προηγουμένως ότι θα επιτύχουμε στους φιλόδοξους κλιματικούς μας στόχους μόνο εφόσον παράσχουμε υποστήριξη σε αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο και θα εξασφαλίσουμε καλή διαχείριση της διαδικασίας προσαρμογής και μετάβασης χωρίς να αφήνουμε κανένα πίσω. Ιδρύματα όπως ε, η ΕΤΕΠ ε, που δημιουργήθηκαν για να προωθούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη, η κοινωνική διάσταση για μας είναι πολύ σημαντική. Και γι' αυτό θα είμαστε βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την εφαρμογή του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης που πρόσφατα παρουσιάστηκε. Θα κοινοτοποιήσουμε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ε, για να ευνοήσουμε τους πολίτες και τους εργαζόμενους στις περιοχές που εξαρτώνται περισσότερο από ορυκτά καύσιμα είναι κάτι που έχουμε κάνει εδώ και καιρό με τις επενδύσεις μας προκειμένου να βοηθήσουμε την ε, οικονομική αναδιάρθρωση ε, περιοχών που εξαρτώνταν από τον άνθρακα. Η ΕΤΕΠ ε, και το Ταμείο μας δεν ε, έχει φυστεί προσπαθειών για να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θα συνεργαστούμε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη και άλλου εταίρου για να αναβαθμίσουμε τι επενδύσει μα και να στηρίξουμε τη δίκαιη μετάβαση προ ένα μέλλον ανθεκτικό για το κλίμα και με απαλλαγμένο ε, από τον άνθρακα. Και θα συμβάλλουμε στις προσπάθειες μετριασμού των κλιματικών αλλαγών. Η μετάβαση φυσικά θα είναι δαπανηρή, αλλά το κόστο τη αδράνεια και το τίμημα τη αδράνειας είναι πολύ μεγαλύτερο. Και παρά τι προκλήσει, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτέ οι επενδύσει περιέχουν και ευκαιρίες και μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ιστορική στιγμή και να υλοποιήσουμε τη μετάβαση εξυγχρονίζοντα τι οικονομίε μα και καθιστώντα τι πιο βιώσιμε και αηφόρε. Και θέλουμε να υπολογίσουμε και στην ε, ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ναβάρο. Ακούσαμε τρεις ομιλητές. Ευχαριστώ τον ε, Αντιπρόεδρο Ρέινερ. Κύριε Μιλόσεβιτς, κύριε συνάδελφε, ε, ελάτε για να μην είμαι και μόνη μου στο Προεδρείο και περνούμε στην πιο διαδραστική περίοδο ανταλλαγής απόψεων σήμερα το πρωί. Όλοι γνωρίζουμε τον κύριο Μιλόσεβιτς, πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κροατικού Κοινοβουλίου. Θα συμπροεδρεύσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Ελπίζω ότι θα λάβετε όλοι τον λόγο. Δίνω τον λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος θα ξεκινήσει τη συζήτηση του Ζακ Φράγκ. Ο κύριο Καμφά. Ευχαριστώ και επιτρέψτε μου να μιλήσω γαλλικά. Χαίρομαι για το σε ακούσαμε. Άκουσα πολύ προσεκτικά τους ομιλητές. Ε, σε δύο-τρία λεπτά θέλω να ανακεφαλαιώσω πού βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την Πράσινη Συμφωνία. Θεωρούμε κατά μεγάλη πλειοψηφία ότι η πράσινη συμφωνία πρέπει να είναι αξιόπιστη και δίκαιη. Αξιόπιστη σημαίνει αξιόπιστη χρηματοπιστωτικά πρώτα απ' όλα. Υποστηρίξαμε με μεγάλη πλειοψηφία και πάλι την μετατροπή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε τράπεζα για το κλίμα. Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν δεδομένη για αυτήν την μετάβαση. Επίσης, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να κάνουμε αυτό το οποίο είπε η κυρία Ναβάρο. Δηλαδή, να προβούμε σε μια ταξινόμηση. Καταστρώσαμε μια, αν θέλετε, ευρωπαϊκή γραμματική για την χρηματοπιστωτική δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όχι μόνο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και εναντί των κεντρικών ευρωπαϊκών τραπεζών και των άλλων συστημικών τραπεζών. Αξιοπιστία σημαίνει επίση αξιοπιστία όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, που είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πιέζουμε λοιπόν για περισσότερου ιδίου πόρου, πράσινου, για την υποστήριξη τη μετάβαση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέρο αυτή τη αξιοπιστία, τη πράσινη συμφωνία, έχει μια χρηματοπιστωτική, χρηματοοικονομική πτυχή έχουμε πιστεί ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε όλε τι μεγάλε πολιτικέ ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ την κατεύθυνση αυτή. Αξιοπιστία επίση σημαίνει ε, αξιοπιστία στον βιομηχανικό τομέα. Γιατί μπορεί να καταστρώνουμε σχέδια, να θέτουμε στόχου, ουδετερό ισοζύγιο το 2050, να βάζουμε όλο και πιο αυστηρού στόχου. Αλλά εάν δεν ακολουθήσει η βιομηχανία με βάση μια κλίμακα αξιών, τότε όλοι αυτοί οι στόχοι θα μείνουν στα χαρτιά. Γι' αυτό και προσπαθούμε σήμερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάστρωση μιας βιομηχανικής πολιτικής. Δηλαδή τι σημαίνει μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση, ουδέτερη όσον αφορά το ισοζυγείο άνθρακο. Τι σημαίνει αυτό για την αυτοκίνητο βιομηχανία, για το χάλιβα, τον άνθρακα και ούτω καθεξής τις βιομηχανίες στις οποίες είμαστε πρωταγωνιστές και βεβαίως θέλουμε να συνεχίσουν να είμαστε πρωταγωνιστές. Συνεχίζουμε επίσης να προσπαθούμε να καταστρώσουμε ένα μηχανισμό ελέγχου του συζυγίου άνθρακα στα σύνορα. Το οποίο σημαίνει ότι εάν αυξηθούν οι τιμές του άνθρακα, των μετάλλων αυξηθούν, κάτι το οποίο θα γίνει, φαίνεται ήδη αυτό, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει κάποιος μηχανισμός να εξασφαλίζει ισότιμη εφαρμογή των κανόνων για τους Ευρωπαίους για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες για να μην ε, χρειαστεί να φύγουν θέσει εργασίας από την Ευρώπη. Αξιοπιστία λοιπόν στον βιομηχανικό τομέα, αξιοπιστία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Και τέλος, το δίκαιο του πράγματος. Κύριε Ρέντερ, έχετε δίκιο. Χρειαζόμαστε έναν δίκαιο μηχανισμό μετάβασης. Αν δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό, θα το δημιουργήσουμε επειδή το ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμό αυτό είναι γέννημα θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι στόχοι είναι δύο προκειμένου. Μια κοινωνική δικαιοσύνη και μια γεωγραφική δικαιοσύνη για τι περιφέρειε. Να μην ξεχάσουμε λοιπόν ποιε περιφέρειε μα χρειάζονται περισσότερο. Και αυτό πρέπει να πάρει τη μορφή δεσμεύσεων. Δηλαδή, όχι μόνο επιδοτήσει, όχι μόνο κονδύλια τα οποία πέφτουν με λέξη χωρί συγκεκριμένο στόχο πρέπει να συνδέονται με ένα τοπικό, περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Και αυτή είναι και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, περισσότερα με κονδύλια, δεσμεύσεις δε, για την κινητοποίηση των επενδύσεων στην ενεργειακή μετάβαση, στον ηλεκτρισμό, στην πράσινη χημική βιομηχανία και ούτω καθεξής, εκεί που χρειάζεται, στις περιφέρειες που χρειάζεται. Και υπάρχουν και άλλες ε, διαστάσεις που δεν πρέπει να ξεχάσουμε αλλά δεν έχω χρόνο το λέω όμως στους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων το λέω στις χώρες που αισθάνονται ότι πλήττονται από τη μετάβαση λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στο πλευρό σας για να γίνει η μετάβαση αξιόπιστη με τρόπο επιστημονικό, με βάση επιστημονικά δεδομένα, αλλά και να είναι αξιόπιστη, όπως είπα, και στον βιομηχανικό τομέα. Διότι δεν θέλουμε να διαλέξουμε μεταξύ βιομηχανία και κλίματο. Όχι, θέλω να είμαστε δίκαιοι και έναντι των περιφερειών, διότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια Ευρώπη η οποία αφενό κατά ένα μέρο τη θα οδεύει προ προς το ενεργειακό, το ενεργειακό ισοζύγιο και άλλοι να ακολουθούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Και τώρα θα ακούσουμε μιλητέ από από το, ε, από τα κοινοβούλια, το, κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια. Με βάση αυτήν την κάρτα, ε, ο κύριος Μιχαήλ Μπαχ ε, είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην Ευρώπη Θέλουμε να είμαστε ηγέτες, ε, το ίδιο ισχύει και για τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Όμως ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, με στόχους που δεν μπορούμε να πετύχουμε για το 2050. Ε, δεν θα πρέπει να απαιτούμε υπερβολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει πολλές φορές, γι' αυτό αντί για μεγάλα λόγια για την κλιματική ουδετερότητα στην Ευρώπη, σε εθνικό επίπεδο να προσπαθήσουμε να δραστηριοποιηθούμε. Σίγουρα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και επίσης πρέπει να έχουμε κατά νου και το κόστος ε, για την μετατροπή. Γιατί για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις ε, θα προκύψουν επιβαρύνσεις ε, τις οποίες ε, θα πρέπει κάπως να καλύψουμε, να κάνουμε περικοπές σε άλλους τομείς. Αν δεν το κάνουμε αυτό η κοινωνία μας θα διαλυθεί. Βεβαίως θα υπάρχουν νικητές αλλά θα υπάρχουν και οι τιμένοι. Και αυτό πρέπει να το πούμε ειλικρινά στους ανθρώπους. Εμείς στη Γερμανία ακολουθούμε ένα δύσκολο δρόμο. Προσπαθούμε να απομακρυνθούμε από την πυρηνική ενέργεια και από τον άνθρακα η κυρία Μέρκελ Μέρκελ ε, είπε ότι μέχρι το 2030 θα έχουν περιοριστεί εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα κατά 50% ε, με δικά μας χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και για μια βιομηχανική χώρα αυτό είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές βεβαίως και πρέπει να συμβάλλουν προς την επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά θέλω να σας προειδοποιήσω, να σας πω ότι για μέτρα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή ε, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες άλλες ε, περικοπές ε, θα πρέπει να υπάρχει πολύ αυστηρή, να υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για τις αγορές γιατί οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να γίνονται μόνο με βάση το πράσινο κριτήριο αυτό θα ήταν σίγουρα κίνδυνος για την σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και για την δυνατότητα ανάπτυξης νέων καινοτομιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, κυρία Τιλιέ από τη Γαλλία. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι σήμερα υπάρχει μια επιστημονική συνένεση, αλλά και συνένεση μεταξύ μα για την κατεπίγουσα ανάγκη να επιταχύνουμε τι προσπάθειέ μα για να καταπολεμήσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ. Επίσης, θα πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι σήμερα πιο σημαντικό, γιατί έχουμε μια τεράστια πρόκληση μπροστά μας. Ε, κάτι που προϋποθέτει τεράστιες επενδύσεις, αλλά και σκέψη ως προς τη μέθοδο. Ο Πασκάλ Καμφά πολύ σωστά το επισήμανε. Θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Χρειαζόμαστε και χρηματοοικονομική αξιοπιστία, αλλά και βιομηχανική αξιοπιστία. Ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη και μια νομοθετική αξιοπιστία, γιατί εμείς νομοθέτες είμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και να αναλύσουμε και τη μέθοδο. Δεν, δεν θα πρέπει να ακολουθούμε παράλληλες πορείες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε σε όλα τα σχέδια που εγκρίνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε δύο παράλληλες πορείες που δεν συναντιόνται. Θα πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε την ενεργειακή μετάβαση και πώς θα καταπολεμήσουμε τα κλιματικά μας προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω έκκληση σε όλους να σκεφτούμε διεξοδικά τη μέθοδο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα επίση να σα επισημάνω, αν έχετε συγκεκριμένη ερώτηση προ καλεσμένου μα, να το επισημάνετε. Ο κύριο Πόπ έχει το λόγο από τη Ρουμανία. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ και ε, Εθνική Βουλευτέ, νομίζω ότι όλοι εστερνιζόμαστε τι φιλοδοξίε Ευρωπαϊκή Ένωση για τι κλιματικέ αλλαγέ. Δαψιλή χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθούν οι προτεραιότητε τη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Επίσης κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να επηρεάσει τα διαρθρωτικά ταμεία και την πολιτική συνοχή. Θα πρέπει να περικοπούν αυτά τα κονδύλια. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση του αντικτύπου σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων για το 2030 και 2050. Ανά κράτος μέλος. Αυτό θα πρέπει να εξαρτήσει ε, να ε, λάβει υπόψη τον εθνικό προπολογισμό και να ληφθεί υπόψη στη χρηματοδότηση. Σίγουρα δεν θα πρέπει να καθυστερούμε, αλλά να μην ξεχνούμε ότι η μετάβαση προς την πράσινη οικονομία προϋποθέτει ιδιαίτερα μέτρα χώρα ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης ε, σε ό,τι αφορά τι κλιματικέ αλλαγέ και μερικά κράτη-μέλη ε, θα απαιτήσουν πολύ μεγαλύτερε επενδύσει υποδομέ και άρα κατάλληλη χρηματοδότηση. Επίση, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το κοινωνικό κόστο και την, τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα. Σίγουρα οι κλιματικέ αλλαγέ δεν έχουν σύνορα. Πώ θα δράσουμε όμω σε εμπορικό επίπεδο σε σχέση με άλλε οικονομίε που δεν θα εφαρμόσουν αντίστοιχε δράσει για το κλίμα και το περιβάλλον ή δεν θα ασχοληθούν καθόλου στη δημόσια πολιτική του με τα θέματα αυτά. Σα ευχαριστώ από τη Φιλανδία. Είναι ο επόμενο ομιλητή. Ο κύριο Μπάρτι Άινεν. Σας ευχαριστώ για τη στεντόρια φωνή σα. Ευχαριστώ, ήταν πολύ ενθαρρυντικές οι παρουσιάσει, γιατί φαίνεται ότι αλλάζουν οι συμπεριφορέ. Αλλάζει η συμπεριφορά για να περιλάβουμε περισσότερε αξίε, αλλά έχουμε και περισσότερε προσδοκίε. Γιατί η οικονομία τη αγορά καθοδηγείται από προσδοκίε και η μετάβαση σε μια οικονομία χωρί ορυκτά καύσιμα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί έναν γενικό προσανατολισμό των επενδύσεων. Και φυσικά ε, θα πρέπει να υπολογίζουμε και στην προορατικότητα των επενδυτών. Σίγουρα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα έχει συνέπειες. Αλλά όταν ένας επενδυτής ε, βλέπει το μέλλον ε, και δεν το βλέπει ελκυστικό ε, ή βλέπει ότι περιορίζονται τα ορυκτά καύσιμα ή ενεργοβόρες βιομηχανίες νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε κάπως και τις προσδοκίες και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνάμεις της αγοράς όλους τους ιδιώτες ε, που με τις δράσεις τους μεμονωμένα θα συμβάλλουν στη μετάβαση. Φυσικά όπως είπε και ο κύριος Κάρνη, το TCFD, αυτή η ειδική ομάδα για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες για το κλίμα είναι πολύ σημαντική, αλλά και η ταξινομία το ίδιο, το εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης. Και αυτό είναι σημαντικό για του μεγάλου θεσμικού επενδυτέ, γιατί το χρήμα μιλάει. Και θα επενδύσουν σε ένα μέλλον χωρί ορυκτά καύσιμα, εφόσον είναι ελκυστικό και προσοδοφόρο για αυτού και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει αυτή την αλλαγή στις προσδοκίες. Κατά τη γνώμη μου, ε, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο από την άποψη αυτή θα είναι ένας πανευρωπαϊκός προϋπολογισμός για το διοξίδιο του άνθρακα και τον προσδιορισμό των τιμών δικαιωμάτων εκπομπής και κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει αυτός ο, ο μηχανισμός να επεκταθεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε βαρτάνιαν και η κυρία Σταύρου από την Κύπρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, δράτω με της ευκαιρίας να χαιρετήσω την πρόσφατη δημοσίευση της Πράσινης Συμφωνίας που έχει ως επίκεντρό του τον άνθρωπο και φιλοδοξεί να μας οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου οικολογική μετάβαση συμφωνώ με τις εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες της ένωσης που εφαρμόζουν χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα θα πληγούν εντονότερα από τον οικολογικό μετασχηματισμό. ευελπιστούμε ότι ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης θα παρέχει την απαραίτητη χρηματοδοτική τεχνική και διοικητική στήριξη για διευκόλυνση των κρατών και περιφερειών που πλήττονται εντονότερα από την οικολογική μετάβαση προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των περιβαλλοντικών τους δεσμεύσεων. Η αποτελεσματική διαχείριση και ο μετριασμός του αρνητικού αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής απαιτεί την υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης καθώς και μέτρων εθνικής προσαρμογής περαιτέρω απαιτείται οριζόντιος συντονισμός ανάμεσα σε όλες τις σχετικές πολιτικές Παραδείγματο χάρη γεωργία ενέργεια μεταφορές βιομηχανία τουρισμό υγεία οικονομία περιβάλλον. θα πρέπει να υπάρξουν συνέργειες και συλλογική προσπάθεια ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Κλείνοντα θα ήθελα να τονίσω ότι η παροχή στοχευμένων κινήτρων για την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, για δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών υποδομών και για διευκόλυνση της εφαρμογή των εθνικών δεσμεύσεων για την ενέργεια και το κλίμα, η προώθηση της χρήση της ηλεκτρική ενέργεια και ο περιορισμό των εκπομπών άνθρακα στον τομέα των μεταφορών, η διείσδυση καθαρότερων καυσίμων όπω το φυσικό αέριο στον τομέα τη ενέργεια η βελτίωση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι μερικά από τα μέτρα που συμβάλλουν σημαντικά στον μετριασμό και τη διαχείριση του αρνητικού αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, Πολωνία. Ο κύριος Αξιότιμοι συνάδελφοι, κύριοι Συμπρόεδρε, αγαπητά μέλη της ε, συνέλευσης, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι πολύ ωραία προπτική και οι Πολωνοί προσβλέπουν σε αυτή την υλοποίηση. Βέβαια σήμερα επικεντρωνόμαστε στην κλιματική πολιτική που είναι πολύ σημαντική εν ώψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο ρόλος όμως του άνθρακα ε, δεν είναι ένα μικρό τμήμα αυτής της συζήτησης. Οι σημερινές τεχνολογίες ε, και το φυσικό αέριο είναι 15-18% μείωση των ε, εκπομπών σε σχέση με τον άνθρακα. Και αυτή η προοπτική προκαλεί χώρες όπως η Πολωνία ε, να υιοθετήσουν στόχους που ξεπερνούν τις οικονομικές και δημοσιονομικές τους ε, ε, δυνατότητες ακόμη και με δανεισμό με ευνοϊκούς όρους έχουμε τεράστιες δαπάνες αλλά και από και από η ιστορική άποψη. Είχαμε για 50 χρόνια καθυστέρηση μετά την παραμονή μας τόσα χρόνια από τον ρωσικό ζυγό. Οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά στο βαθμό ανάπτυξη των χωρών και την ε, δυνατότητα αναδιάρθρωσης. Εμεί θα πρέπει να αναδιαρθρώσουμε τα τρία τέταρτα τη παραγωγή ενέργεια ε, στην παραγωγή μα. Και 7,5 δισεκατομμύρια ε, στο Ταμείο Δίκαιη Ανάπτυξη είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τι δαπάνε που χρειαζόμαστε. Θέλουμε να αισθενιστούμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά με τι οικονομικέ και κοινωνικέ μα συνθήκε μπορούμε να πούμε σήμερα ότι μόνο στο δεύτερο μισό του αιώνα θα είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε αυτή τη νέα πράσινη συμφωνία. Έχουμε ήδη κλείσει 30 ανθρακοριχεία στην Πολωνία λόγω έλλειψης κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και έχουμε πολλά ανθρακοριχεία που ε, ετοιμάζονται να κλείσουν. Έχουμε ε, ο 8.000 θέσει απασχόληση που έχουμε χάσει λόγω του κλεισίματο αυτών των αθρακοριχείων. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι συνέπειε. Οπότε, τι προοπτικέ υπάρχουν για τη δική μα μετάβαση. Χρειάζονται τεράστιε επενδύσει, ε, τεράστιε δαπάνε για τη μετάβαση αυτή. Και ο ρυθμό μα θα πρέπει να εξαρτηθεί από τι δυνατότητέ μα. Και επίσης, 500 ε, εκατομμύρια είναι το κόστος ε, για την αναδιάρθρωση ενός και μόνο αθρακοριχείου. Και σκεφτείτε πόσα έχουμε εμεί που θα πρέπει να αναδιορθώσουμε. με τι ρυθμό θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε όλα αυτά τα βήματα. Είναι πολύ δύσκολο θέμα. Ήδη έχουμε αναλάβει πολλέ προσπάθειε και έχουμε κάνει πολλέ δράσει, αλλά η πραγματικότητα μα έχει δείξει ότι είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτέ τι φιλόδοξε πολιτικέ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Τούσεκ από την Κροατία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών ε, γίνονται αισθητέ ε, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και γι' αυτό ε, και η, αντιμετώπιση του κλίματος είναι ύψιστη πολιτική προτεραιότητα. Οι αλλαγές στην συλλογική μας συμπεριφορά γίνονται με πολύ αργό ρυθμό. Και επίσης θα πρέπει να μιλούμε για ολοκληρωμένες ε, κατευθυντήριες γραμμές, ε, διατομιακές πολιτικές που δεν θα αφήνουν κανένα πίσω. Επίσης θα πρέπει να επενδύσουμε σε καινοτομία, σε πράσινες φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες και να μην ξεχνούμε ότι έχουμε ενιαία αγορά που θα πρέπει να είναι όλο και πιο πράσινη και φιλοπεριβαλλοντική. Και θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις και οι τομείς να λάβουν υπόψη κάποια πράσινα μέτρα. Και αυτό να το λάβουμε υπόψη και στις ε, δημόσιες ε, συμβάσεις για να έχουμε ε, βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και μια αποτελεσματική οικονομία. Σημαντικό, σημαντική πρόκληση στον δρόμο τη ε, κλιματική ουδετερότητα είναι η εξασφάλιση της, ε, του ενεργειακού μα αναφοδιασμού. Εμεί στην Κροατία έχουμε μεγάλο ενεργειακό δυναμικό λόγω τη εξαιρετική μα θέση ε, και τη δυνατότητα μέγιστη αξιοποίηση τη ηλιακή ενέργεια που είναι η φθηνότερη πηγή ανανεώσιμη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν έχουν όλε οι χώρε το ίδιο δυναμικό. Θα πρέπει λοιπόν ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξη και το δυναμικό, να προσπαθήσει κάτι ε, χώρα με το ρυθμό της να, να προσαρμοστεί στις κλιματικές αλλαγές και να μην εξαρτάται από ορυκτά καύσιμα. Εμείς στη διάρκεια της Προεδρίας μας ε, θα λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μεμονωμένων περιοχών. Επίσης, ε, έχουμε πει ότι για την επόμενη δεκαετία θα χρειαστεί ένα, ένα τρισεκατομμύριο ευρώ επενδύσεις. Οπότε οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2021-2027 θα έχουν κέριο ρόλο. Θα πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συμβιβασμούς, αλλά όχι εις βάρος σημαντικών κονδυλίων όπως είναι αυτών της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Και επιστρέφω στους ομιλητές. Δεν υπήρχαν ερωτήσεις, αλλά ο κ. Κάρνη όσον αφορά τα δημοσιονομικά και τελευταία παρατηρήση. Είπε και κάτι σχετικό ο πλονός συνάδελφος ε, σχετικά με τα δισεκατομμύρια τα οποία πετούνται για την μετάβαση προκειμένου. Κάρνε, θέλω να διτυπώσω λοιπόν τέσσερις σκέψεις. Πρώτον, για τον κύριο Καφέ, και ε, προς τον Ρουμάνο, σαν ο σχολίασε τι γίνεται με τις χώρες που δεν ακολουθούν εν ώψη της COP26 και τι γίνεται με τις εκπομπές κατηγορίας 3. Αυτές ε, συμπεριλαμβάνονται φυσικά στους πολιτισμούς και όσο περισσότερο συμμετέχουν μικρότερες εταιρείε στους πολιτισμού, τόσο περισσότερες χώρες και επιχειρήσεις ακολουθούν. Δηλαδή αυτό είναι ο θετικός τρόπος της προσαρμογής της μετάβασης. Πρέπει φυσικά το άρθρο 6 της διαδικασίας ΚΟΠ να το δούμε καλύτερα σχετικά με την αντιστάθμιση, την διασυνοριακή αντιστάθμιση δικαιωμάτων έτσι ώστε να αποφεληθούν όλοι με τρόπο ισότιμο. Και σίγουρα οι φορεί, οι δεσμοί μάλλον ε, προκειμένου μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν. Πάντως πριν φτάσουμε στις, ε, στα αρνητικά μέτρα υπάρχουν θετικά. Και τέλος, επειδή είπατε υπάρχει υπεπερασμένος προπολογισμό, δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω για τις τάξεις μεγέθους θα ενισχύσω όμως αυτό το οποίο είπε η κυρία Νεβάρο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ότι αυτή είναι η πιο αποδοτική τρόπη να αξιοποιήσουμε τα δημοσία κονδύλια γιατί έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, έχουμε μόχλευση. Επίσης έχουμε και εγγυήσει από την Πράσινη Συμφωνία που είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο και το οποίο κάτι κάνει και για τη διαχείριση κινδύνων από το κλίμα, από τη μεταβολή του κλίματος. Το οποίο συνάδει με αυτό το οποίο είπε ο Φιλανδός συνάδελφος. Ναι και στην καινοτομία, σύμφωνα απολύτως, ο κόσμος περιμένει μια θετική ατζέντα, μια θετική δυναμική και είμαστε κοντά σε αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε και τις ιδιωτικές αγορές να ακολουθούν. Υπάρχει ήδη μια θετική λοιπόν δυναμική και στην ιδιωτική οικονομία και πιστεύω ότι θα δούμε πιο σημαντικά βήματα. Δεν υποτιμώ καθόλου αυτή την εξέλιξη. Και τέλος, ορισμένοι μιλητές ορθώς τόνισαν, όπως και εσείς, την αξία, τη σημασία της δίκαιης μετάβασης. Οι στόχοι τη μεγάλη επιχειρήση σαφώ βοηθούν, ιδιαίτερα να βάλουμε μέσα και την κατηγορία 3, εκπομπές εκπομπέ κατηγορία αλλά εδώ έχουμε και τον ρόλο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων που θα σχεδιάσουν του μηχανισμού, του σχετικού μηχανισμού για την παροχή επανεκπαίδευση μεταξύ άλλων και ούτω καθεξής. Και τέλος, τέλος σύμφωνα με τον Guy Ryder ο οποίο είπε ότι χωρίς την κοινωνική δικαιοσύνη και χωρίς την δίκαιη μετάβαση υπονομεύουμε κατά τα άλλα εξαιρετικές πολιτικές. Ευχαριστώ. Κύριε Ράιντερ, λέει πρόεδρο. Είπατε γενικητέ και χαμένου στην αρχή. Τι γίνεται με του εργαζομένου. Γιατί ο κόσμο, ναι, η κοινή γνώμη τουλάχιστον λέει ναι στην δράση για το κλίμα, αλλά στην πράξη τι θα σημαίνει αυτό για τι δουλειέ. Είπα με παραδό στην πρωτολογία μου ότι ο διάλογος, η συζήτηση αφορά πλέον άμεσα και τον χώρο της εργασίας. Λοιπόν, δεν εκπροσωπώ ούτε του μεν, ούτε του του εργοδότε, ούτε του εργαζόμενου. Αλλά θα μπορούσε να πει ένα παρατηρητή ότι με μεγάλη ταχύτητα καταφέρουμε να πετύχουμε παγκοσμίω συνένεση όσον αφορά το κόστος. Δηλαδή, το που θα πάει η εργασία και πώς θα συγκεραστεί το δική μας εργασία με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Δεν υπάρχει καμία εμφιβολία ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο, πολύ εγχείρημα έτσι, και εξαιρετικά φιλόδοξο. Λοιπόν, αυτό το οποίο προκύπτει από την συζήτηση είναι, είναι και αυτό. Πόσο πολυσύνθετο είναι το εγχείρημα. Και είπαν πολύ αξιοπιστία. Ναι, χρειαζόμαστε χρηματοπιστωτική αξιοπιστία. Αυτό συζητούμε σήμερα μεταξύ άλλων και αυτό αφορά τον ιδιωτικό τομέα και τις δημόσιες επενδύσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια δοκιμή, αν θέλετε, αξιοπιστίας και δικαιοσύνης ταυτόχρονα, για να μην έχουμε μόνο χαμένους. Ε, χαμένοι θα υπάρχουν σίγουρα στην πρώτη φάση, αλλά δεν θέλουμε να είναι ιτημένοι και στο τέλος. Αυτό δεν θα είναι δίκαιο. Γι' αυτό λέω αξιοπιστία και δικαιοσύνη. Και προ τον πρόεδρο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο υπάρχει θέμα βιομηχανική αξιοπιστία. Διότι αυτή τη στιγμή η βιομηχανική υποδομή αλλάζει, η εργασία αλλάζει και γι' αυτό περισσότερο από οπουδήποτε αλλού τα θέματα του κοινωνικού διαλόγου εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να συζητηθούν με τη συμμετοχή των εργαζομένων και να θεωρηθούν θέματα προτεραιότητας. Στον Χάλιβα, στον Άνθρακα, οι επιχειρήσει, ε, οι εργαζόμενοι ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει και μπορούν να συμβάνουν στον διάλογο. Και έτσι προχωράει η Ευρώπη με συνένεση. Αυτό είναι ο ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα. Και τέλο, πάλι για την αξιοπιστία, όπω είπε και ο κ. Σκαρνή και όπω είπε και ο Φιλανδός βουλευτής. Ναι, πρέπει να διχειριστούμε τις προσδοκίες, τις προσδοκίες των αγορών, ώστε επενδυτέ οι αγορές να έχουν κατεύθυνση, αλλά να διχειριστούμε και τις προσδοκίες των πολιτών που περιμένουν πολλά από εμάς. Γιατί εν τέλει εκεί θα θεμελιώσουμε και την πολιτική μας νομιμοποίηση στους πολίτες. Ανησυχώ πρέπει να πω κατά υπό την έννοια ότι τίθενται εύλογα ερωτήματα. Τι είναι αυτή η πράσινη συμφωνία και πώς συγκεράζεται με άλλους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δημοσιονομικά, τα φορολογικά και ούτω καθεξής. Πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά μαζί. Θα ήταν προβληματικό εάν η πράσινη συμφωνία γίνεται αντιληπτή ως μια αντίφαση που υπονομεύει τους άλλους στόχους. Όχι, η πράσινη συμφωνία είναι αναπτυξιακή συμφωνία. Δεν είναι απλώς ένα προσάρτημα στις άλλες πολιτικές. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ναβάρο, για τη χρηματοδότηση και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για τη στήριξη τέτοιων επενδύσεων φιλοπεριβαλλοντικών. Όπως σας είπα, είμαστε η τράπεζα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη βάζουν κεφάλαιο στην ΕΤΕΠ και με το κεφάλαιο αυτό μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε στην αγορά και να χρηματοδοτήσουμε στη συνέχεια επενδύσεις που είναι κρίσιμες για την βιωσιμότητα της Ευρώπης και για την οικονομική ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά θα πρέπει να εστιαστούμε στην μετάβαση και θα πρέπει να στηρίξουμε τη δίκαιη μετάβαση, οπωσδήποτε. Αλλά σε τελική ανάλυση μιλούμε για μια διαδικασία εξυγχρονισμού. Και αν κάνουμε αυτό το μετασχηματισμό με λάθος τρόπο, αυτοί που ε, θα πληγούν περισσότερο δεν θα μπορέσουν να μετριάσουν αυτές τις αρνητικές συνέπειες. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε για να διαχειριστούμε σωστά τη μετάβαση και με τρόπο ώστε όλες οι περιφέρειες να υποφεληθούν από τη διαδικασία εξυγχρονισμού. Επίσης και η κλιματική διπλωματία θα είναι σημαντική αυτή τη στιγμή γιατί η Ευρώπη χρειάζεται να προσετεριστεί και άλλες χώρες, τρίτες χώρες. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει ήδη υποστήριξη από πολλές χώρες και από κάποιες δικαιοδοσίες που ίσως δεν ακούγονται τόσο ηχηρά αλλά έχουν περιφέρειες και έχουν πολίτες που επίσης ασκούν πιέσεις και ζητούν αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Γιατί οι πολίτες ενδιαφέρονται και ανησυχούν. Και στην Ευρώπη έχουμε την κοινωνική διάσταση, αλλά τέτοια κοινωνική διάσταση υπάρχει και εκτός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρώπη. και θα πρέπει να τη στηρίζουμε, όπως κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο μεγαλύτερος δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες για να, να τις διευκολύνουμε στη δική τους μετάβαση. Γιατί η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και το κλίμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Τώρα να δώσω το λόγο στον συμπρόεδρο, τον Ντομαγκόη Μιλόσεβιτς, για να συντονίσει το δεύτερο γύρο της συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην Κύπρο τώρα, τον κύριο Βότση. Okay. Υπό το φως της επικείμενης οριστικής αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή τον Νοέμβριο του 2020, θα ήθελα να εκφράσω τις έντονες ανησυχίες μου ω προ τον κίνδυνο που ελοχεύει για απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συνεπία τη υποχρέωση συμμόρφωσή του με υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα που συνεπάγονται αύξηση του κόστου παραγωγή. Οι διεθνεί εταίροι δεν δεσμεύονται από του φιλόδοξου στόχου που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Αναμφίβολα, η εφαρμογή υψηλότερων περιβαλλοντικών προτύπων και οι βιώσιμε έξυπνε επενδύσει εγγυώνται την αναβάθμιση του ιδιωτικού επίπεδου και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Παράλληλα όμω, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το κόστο που συνεπάγεται η συμμόρφωση με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει δεν θα λειτουργήσει ανασταλτικά ω προ την οικονομική του βιωσιμότητα και δεν θα οδηγήσει σε μεταφορά των παραγωγικών μονάδων των επιχειρήσεων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω χαμηλότερου κόστου παραγωγή. Περαιτέρω, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη εντελεχού επανεξέταση των οικονομικών και κοινωνικών πτυχών τη Πράσινη Συμφωνία, καθώ και εκπόνησης εκθέσεων αντικτύπου σε κάθε χώρα ξεχωριστά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο οικολογικό μετασχηματισμό είναι δίκαιο και χωρί αποκλεισμού. Η ευθυγράμμιση των οικονομικών πτυχών τη Πράσινη Συμφωνία με του υπόλοιπου στόχου μακροοικονομική σταθερότητα αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα κράτη-μέλη τη Ένωση στην ολότητά του. Καταλήγοντα, θα ήθελα να τονίσω ότι οι πρόνοιε τη Πράσινη Συμφωνία είναι αδύνατο να ελοπιθούν εν μία νυχτή, δεδομένου ότι ο οικολογικό μετασχηματισμό απαιτεί πρώτη στα ριζική αλλαγή νοοτροπιών, ώστε η μετάβαση να είναι ομαλή και ανώδυνη για του πολίτε και τι επιχειρήσει επειδή ζητήσατε ερώτηση πώς σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που θα προκύψουν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που δεν υιοθετούν τους δικούς μας φιλόδοξους στόχους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο Λουξεμβούργο τώρα. Ο κύριος Μάρκ. Euh- Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ομιλητές για τις εξαιρετικά φιλοδοξές ομιλίες τους. Συμφωνώ. Ε, το ρέτημα μου με αυτό όμως ακριβώς συναρτάται. Εργάζομαι στο Λουξεμβούργο ε, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, ε, με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, ε, ο κ. Κάρνε είναι ένας από αυτούς. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη λοιπόν, απόσταση και εξηγούμε. Επέστρεψα στο Λουξεμβούργο και διαπίστωσα ότι ο κόσμος δεν συμφωνεί όσον αφορά το κατεπήγον του θέματος, την ανάγκη κατεπήγουσες δράσης. δηλαδή. Συνεχίζουμε όλοι ε, επί της πεπατημένης και δεν ξέρω αν ο κόσμος ξέρει, βολευόμαστε όλοι με την πεπατημένη αντί να αλλάξουμε τον ε, τρόπο δράσης μας γενικά. Ε, μιλήσατε για την TCFT, κανείς δεν την ξέρει. Και φοβούμε ότι πέραν της κατονιδής ανθρώπινης αντίσταση στην αλλαγή υπάρχει αντίσταση και στο επίπεδο των διοικήσεων, των κυβερνήσεων. Δεν γνωρίζουν ε, δεν έχουν διαπιστώσει αυτό που διαπιστώνουμε. Και, κύριε Κάρνη, θα μπορούσατε να με διαβεβαιώσετε ότι εξαιρετικοί διοικητές των κεντρικών τραπεζών δεν είναι σκεπτικιστές όσον αφορά τη μεταβολή του κλίματος. Με ποιους είναι οι κεντρικοί τραπεζίτες. Θα υιοθετήσουν μια πολιτική από την κορυφή προς τη βάση που θα αφορά τον κόσμο, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού υπάρχει πλειοψηφία μεταξύ της κοινή γνώμη όσον αφορά την αποδοχή της μεταβολής του κλίματος. Λοιπόν, που πηγαίνουν οι πολιτικές μας. Φοβούμαι ότι εμείς χαράσουμε πολιτικές, υπάρχει όμως στη βάση πολύ μεγάλη αντίσταση στην αλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Μικαλεφ από τη Μάλτα. Πρόεδρε, αύριο το Συμβούλιο θα προγραμματίσει πώς ακριβώς θα επενδυθούν τα κονδύλια μας κατά επόμενα 7 έτη, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές μας, πώς θα κατορθώσουμε να έχουμε πλεονεκτήματα, πώς θα επωφεληθεί κάθε κράτος μέλος. Αν δεν όλα αυτά ε, θα υπάρχει πρόβλημα με την ευρωπαϊκή πολιτική. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κανείς ε, δεν θα παραμείνει πίσω μόνος του σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια δίκαιη οικονομική και κοινωνική πολιτική. Η ε, ποικιλομορφία μας βοηθάει έτσι ώστε να κατανοήσουμε τους ευέλικτους μηχανισμούς και για να μπορέσουμε να επιτύχουμε πετύχουμε τους στόχους μας ε, χωρίς να δημιουργούμε ε, συστήματα που δεν βοηθούν. Όπως είπε και ο πρόεδρος ε, κύριος Σασόλη, πολλά κράτη-μέλη σκέπτονται δυστυχώς μόνο τη δική τους τη χώρα και όχι την Ευρώπη. Καλό που ακούμε εμπειρογνώμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μας ομιλούν, μας απευθύνουν το λόγο αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου και τις γειτονές μας. Να μην ξεχνάμε ότι τα μικρά κράτη θα επηρεαστούν πολύ περισσότερο. Η Μάλτα, παραδείγματο χάρη, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και ας μην ξεχνάμε, ο ευρωπαϊκός χάρτης θα αλλάξει ε, γνωρίζουμε ότι ακραίες ε, καιρικές ε, συνθήκες θα επιτείνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πολλά κράτη-μέλη ε, δεν έχουν οικονομίες ε, κλίμακας. Γι' αυτό λοιπόν ας μην ξεχνάμε ότι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας μπορούν να αγκάσουν ορισμένες χώρες ε, να παραμείνουν πιο πίσω. Γι' αυτό, ναι, μεν η ηγετική θέση, αλλά μην ξεχνάμε ότι και κάθε χώρα είναι διαφορετική. Ξεκινάμε από εδώ, απευθυνόμαστε στα Εθνικά Κοινοβούλια. Να μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι μία Επίρρος, αλλά και να μην ξεχνάμε τις ε, εθνικές ιδιαιτερότητες. Βεβαίως και είναι σύμφωνη η Πράσινη Συμφωνία, αλλά οφείλουμε να έχουμε και μία ε, κοινωνική και δίκαιη πρόοδο. Θεωρούμε ότι όλες αυτές οι αλλαγές ε, θα ε, λειτουργήσουν ως καταλήτης ε, στη ζωή μας, να μην έχουμε μόνο κατά νου το κλίμα, αλλά και το πώς προσεγγίζουμε τα πράγματα. Ε, μιλήστε λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Η κυρία Κρετού από τη Ρωμανία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να επαναλάβω κάποια πράγματα για να επιτύχουμε πλειοψηφία. Οι στόχοι μας ε, είναι πολύ σοφοί, η πράσινη σοφία. Δεν είναι ένα είδος ε, εταιρεία που κάνει διαφήμιση για το κλίμα και την πράσινη ενέργεια σε αντιπαραβολή και αντίθεση με την ρηπαίνουσα οικονομία. Η συμπεριφορά ε, η διοίκηση. Ε, εδώ η Πράσινη Συμφωνία δεν μπορεί να είναι μόνο ε, καλές προθέσεις ε, οι ανατολικέ χώρε δεν ξεχνάνε πόσο δύσκολο ήταν να πάνε από την κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία στην ελεύθερη οικονομία, κλείσιμο εταιριών, απώλεια θέσεων απασχόληση. Στη δική μου τη χώρα, τη Ρουμανία, 4-5 εκατομμύρια περίπου εγκατέλειψαν τη χώρα για αυτόν τον λόγο και πήγαν στο εξωτερικό. Στο δυτικό κομμάτι της Ευρώπης, ε, ούτε και εκεί οι εργάτες και οι εργαζόμενοι προστατεύτηκαν λόγω του νεοφιλελευθερισμού. Ε, και πολλοί πήγαν σε χώρες με χαμηλότερους μισθούς. Brexit το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, οι ανισότητες. Όλα αυτά είναι στενά συνδεδεμένα με τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται μόνο για το χρήμα. Μια νέα μεταρρύθμιση θα καταστήσει τους πολίτες ιδιαίτερα ευαίσθητους και δεν νομίζω ότι θα ε, στηρίξουν κάτι που δεν είναι δίκαιο. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας με το 1% στον ευρωπαϊκό Πρέπει να απευθυνθούμε στις ε, κυβερνήσεις μας ε, και στις τράπεζες σχετικά με την πολιτική λιτότητας. κίνητρα πρέπει να βρούμε και τέλος ε, θεωρώ ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν θέλουμε και άλλοι να κάνουν τα ίδια, αυτό θα σήμαινε αποτυχία. Κύριε Κρίστοφα από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Κύριε ε, Συμπρόεδρε του, της Συνέλευσης, ε, θα ήθελα να σας απευθύνω χαιρετισμό από την Βοσνιακή Βουλή Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυρες όλο και πιο ακραίων καιρικών συνθήκων και φαινομένων. Είχαμε δασοπυρκαγιές, ε, ε, όχι μόνο στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο. Και οι κλιματικές αλλαγές μεταμορφώνουν τον κόσμο και προκαλούν ανεπανόρθωτες ζημίες στα οικοσυστήματα που έχει, έχουν πληγεί από τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα. Αν είμαστε προετοίμαστοι από τις ε, κλιματικές, στις, απέναντι στις κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουμε αρνητικά και την οικονομία μας. Ε, και οι πυρκαγιές, οι ανοβρίες, οι πλημμύρες πλήττουν την πυρκαγιά. Τη, ε, επιδεινώνουν την οικονομία και από τις πλημμύρες που έχουμε υποστεί πρόσφατα έχουμε διαπιστώσει πώς επηρεάζονται και οι υποδομές και η οικονομία μας από τέτοια καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό και θεωρώ ειδικά σημαντικό να, που βρέθηκε η Βοσνία Αρζεγοβίνη στην ομάδα των χωρών που κύρωσαν τη Συμφωνία των Παρισίων για τις κλιματικές αλλαγές. Εκεί διατρανώνονται πολύ φιλόδοξοι στόχοι και μέτρα για το μετριασμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Και τώρα ε, ως νομοθέτες θα πρέπει να εντείνουμε τις δραστηριότητες και να θεσπίσουμε τις απαραίτητες νομοθετικές διατάξεις ώστε να συμβάλλουμε κι εμείς στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Επίσης χρειάζονται οικονομικές, δημοσιονομικές αλλά και κοινωνικές πολιτικές και να προβλέψουμε περισσότερα κονδύλια στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και να επενδύσουμε στη βιομηχανία και την καινοτομία και στις καθαρές φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην, ε, στην αναδάσωση των ε, περιοχών που έχουν πληγεί από δασοπυρκαγιές και να επενδύσουμε γενικώ σε ε, ποιοτικότερο και υγιέστερο μέλλον. Φυσικά πιστεύουμε ότι καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Εν τη ενώση ισχύς, μόνο μαζί θα, μπορούσα, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, έχοντας κατά νου το γεγονός ότι δυστυχώς οι κλιματικές αλλαγές δεν γνωρίζουν σύνορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μπόριανα. Περνάμε στον κύριο Σουτ τώρα από την Εστονία. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που η συζήτηση που κάναμε είναι ζωηρή και ακούγεται ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι αν θα χρειαστεί μετάβαση, αλλά πώς θα τη διαχειριστούμε αυτή τη μετάβαση και τι μπορούμε συλλογικά να πραγματοποιήσουμε και τι μεμονωμένα κάθε χώρα. Και για την Εστονία η διαχείριση αυτής της μετάβασης αποτελεί μείζωνα πρόκληση. Φυσικά θα χρειαστούν χρήματα, αλλά όπως είπαν και πολλοί προλαλήσαντες, ήδη υπάρχουν αρκετά κονδύλια από την ΕΤΕ, από το Ταμείο Δικής Μετάβασης, με χαμηλά επιτόκια, με ευνοϊκούς όρους και μπορούμε με νομοθετικές διατάξεις αλλά και με βάση τις προτιμήσεις των καταναλωτών να οδηγηθούμε στην πορεία της μετάβασης. Επίσης, ε, έχουμε ευκαιρία για πρόθεση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, γιατί αν είμαστε πρωτοπόροι στη μετάβαση προς μια οικονομία ουδέτερη άνθρακα, θα έχουμε ένα προβάθισμα παγκοσμίω. Γιατί δεν μιλούμε μόνο για τις υφιστάμενες τεχνολογίες που θα μας οδηγήσουν στο στόχο μας, αλλά θα έχουμε και νέες τεχνολογίες. Θα μπορέσουμε να εφεύρουμε νέες τεχνολογίες και συνδυάζοντας παλιές και νέες τεχνολογίες ε, θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Και όσο περισσότερο στρεφόμαστε προς την καινοτομία, ε, στην προσπάθεια μετάβασης ε, τόσο πιο ανταγωνιστική θα γίνουμε παγκοσμίω. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ξεκίνησε ω ε, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Ήρθε η ώρα να γίνουμε η Ένωση των Νέων Τεχνολογικών, Τεχνολογιών συγγνώμη, και της καινοτομία. Η κυρία Σίκουτ από την Εστονία και πάλι. Πρόεδρε, ο ρόλο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε και ο συναδελφό μου μόλι πριν από λίγο, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Συμφωνώ με αυτή την απόφαση. Χρειαζόμαστε όμω και τα εργαλεία υποστήριξη τη καινοτομία και τη πρόοδου προς νέες πράσινες τεχνολογίες, προς την νέα κυκλική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση δεσμεύθηκε να εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα σε όρους απώλειας θέσεων εργασίας, υψηλότερου κόστους ε, ενέργειας κλπ. Όμως, ακόμη πιο σημαντικό είναι, όπως είπε και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και όπως είπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να πετύχουμε το ουδέτερο ισοζύγιο, αλλά αυτό εξαρτάται από καθημερινές αποφάσεις όλων των πολιτών. Μόνο έτσι θα πετύχουμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο. Το ουδέτερο ισοζύγιο λοιπόν δεν είναι κάτι γενικό, αφηρημένο, αποστασιοποιημένο. Όχι, έχει σχέση με την καθημερινή ζωή. Κάθε ένας από εμάς πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Ο Φιλανδός συνάδελφος είπε διαχείριση προσδοκιών των αγορών. Ναι, πράσινες επενδύσεις θα γίνουν μόνο εφόσον πετυχαίνουν την προσδοκόμενη απόδοση. Και τι θα γίνει, όπω είπε ο συνάδελφο, με τι προσδοκίε των πολιτών. Λοιπόν, και τι δύο πρέπει να διαχειριστούμε και το τονίζω αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωή. Πρέπει να αλλάξουμε, να εξασφαλίσουμε μάλλον πολιτική νομιμοποίηση τη μετάβαση. Ο κόσμο πρέπει να κατανοήσει και να αποδεχθεί την ανάγκη αλλαγής. Προκειμένου τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στο να περάσουν στον κόσμο την ανάγκη της αλλαγή με τρόπο κατανοητό. Η διαχείριση λοιπόν των προσδοκιών των πολιτών είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον κατάλληλα ε, εύλογα φιλόδοξο στόχο τον οποίο έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιταλία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως και είναι σωστό να αλλάξουμε το μοντέλο ανάπτυξης, αλλά να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο που να υπηρετούμε την ανάπτυξη. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, πριν και ακόμα από την κινέζικη κρίση. Ε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ε, καλά τα λέμε όλα αυτά, αλλά να προσέξουμε μην προκύψει καμιά ε, χρηματοπιστωτική φούσκα. Ναι, να αλλάξουμε, αλλά με τα πόδια στη γη και με τη μέγιστη προσοχή, με το μάτι στραμμένο Στου στους ανταγωνιστές, στις πραγματικές επενδύσεις, στην προστασία των επιχειρήσεών μας. Μην ε, αυτοτιμωρηθούμε, αυτομαστιγωθούμε. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να βάλω είναι εσείς ε, σε αυτή τη φάση τη μεταβατική τι σκέφτεστε για τα αέρια μεθανίου και αυτό αφορά όχι μόνο τα ελαφρά οχήματα, αλλά και τα μεγαλύτερα. Καλά όλα αυτά, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο. Και στον διάμεσο χρονικό διάστημα τι θα κάνουμε. Παραδείγματο χάνει στην Ιταλία, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στι άλλε χώρε, αλλά στην Ιταλία έχουμε δει πολλοί ε, που απαγορεύουν την χρήση αυτοκινήτων ε, με δίζελ. Ε, δεν ξέρω τώρα αν αυτό έχει νόημα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά τη γεωργία. Το η πρώτη προστασία του περιβάλλοντος ε, γίνεται από τους ίδιους τους ε, γεωργούς. Ποιος ε, φροντίζει τη γη, ποιος φροντίζει τα δάση, τη θάλασσα, είναι η δική μας η Γεωργία και η δική μας η αλληλείς. Ως εκ τούτου για τη γεωργία εκεί θα πρέπει να έχουμε ελάχιστος περιορισμούς γιατί αλλιώς θα, μειώσουμε την προστασία του περιβάλλοντος. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ όλους σας πάρα πολύ και ευχαριστώ ε, που μας ε, δώσατε την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μια τόσο σημαντική συζήτηση. Όχι, έκανα λάθος, με συγχωρείτε. Έχουμε άλλους ε, δύο συναδέλφους, η κυρία Αγκεστάιν από τη Νορβηγία. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Και ευχαριστώ για την οργάνωση αυτής της κοινοβουλευτικής εβδομάδας. Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εργασίες για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που είναι ιδιαίτερος φιλόδοξη και βρήθη προτάσεων που άμεσα ή έμεσα θα επηρεάσουν και την Νορβηγία. Η Νορβηγία ήδη είναι μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών. Παρόλο που ε, η κυβέρνησή μας ε, ε, μετά τη Συμφωνία των Παρισίων αύξησε τη μείωση των εκπομπών κατά 52% ε, μέχρι το 2030 και μάλιστα στη συνέχεια θα υποβάλει και ε, σχέδιο δράση κυβέρνηση προς το Κοινοβούλιο για να υλοποιήσει αυτούς τους στόχους και οι εθνικοί που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές και το περιβάλλον θα συζητηθούν ε, στην Νορβηγική Βουλή με ιδιαίτερη σημασία. Φυσικά είμαστε υπέρ της δίκης μετάβασης που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω και δεν θα αποκλεί κανέναν. Έχουμε φιλοδοξία να μειώσουμε τις εκπομπές μόνο και να μην μειώσουμε την οικονομική ανάπτυξη ούτε την ευημερία των πολιτών. Ευχαριστώ. Και ο τελευταίος αλλά πολύ σημαντικός, ο εκπρόσωπος από την Ουγγαρία, κύριος Βάριο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, Εκπροσωπώ την Ουγγαρία και είμαι ο πρόεδρος τη Επιτροπή Προϋπολογισμών της Ουγγρικής Βουλή. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα για να παρουσιάσω τη θέση μου. Χαιρετίζουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εφόσον ε, θα, δεν θα είναι μονολυθική αλλά θα έχει και τις 50 αποχρώσεις του πρασίνου. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη συμφωνία ότι έχουμε ανάγκη από ένα νέο οικονομικό μοντέλο, αλλά ε, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα δίλημα αν θα υποστηρίξουμε την απασχόληση ή τον πλανήτη. Έχουμε ένα τεράστιο ανθρακοριχείο σε μια περιοχή της Ουγγαρίας με συμμετοχή και της Siemens και εκεί είχαμε μαζικές διαδηλώσεις κατά της επένδυσης αυτής αλλά το δίλημα που ανακύπτει είναι αν θα πρέπει να κάνουμε επιλογή μεταξύ προστασίας του πλανήτη και προστασίας της απασχόλησης. Δεν θέλω όμω να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τέτοιο δίλημα. Θα μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε. Ευχαριστώ. Και Επιτρέψτε μου, για να ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα τη συζήτηση να πω και εγώ λίγα λόγια για το θέμα αυτό. Όλοι ανησυχούμε ιδιαίτερω για το τι πλανήτη θα αφήσουμε στα παιδιά μας στις επερχόμενε γενιές, γιατί έχουμε δραματικές ε, καιρικές συνθήκες παντού στον κόσμο. Και οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν και τις μεταναστευτικές ε, ροές σε πολλές σε, πολλούς, σε πολλές υπήρους και ήδη αλλάζουν το κοινωνικό-οικονομικό τοπίο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μοναδική ευκαιρία αλλά και μοναδική ευθύνη να γίνει παγκόσμιο ηγέτη στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά να γίνουμε ηγέτε και σε θέματα εξυπνολήσεων και των νέων τεχνολογιών που χρειάζονται για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ακούσαμε πολλούς λόγους και επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης και σίγουρα θα πρέπει να επιδιώξουμε διακομματική συμφωνία γιατί το περιβάλλον δεν είναι θέμα αριστεράς ή οικολόγων. Όλοι ανησυχούμε για το μέλλον των παιδιών μας και για τις κλιματικές αλλαγές. ανεβαίνει η στάθμη του νερού και θα ήθελα και τα παιδιά μου αλλά και τα εγγόνια μου να ζουν τις τέσσερις εποχές και να μην τις διαβάζουν για τις τέσσερις εποχές μόνο, για τα, μόνο στα βιβλία. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε σημαντικά ηχέγγυα και από τους σημαντικούς εταίρους μας, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, μετά την ε, αναγγελία της αποχώρησης των ΗΠΑ από την Κλιματική Συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους σημαντικούς και μακροπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους. Επίσης δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε μόνο οι δικέ μας μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή οι δικοί μας πολίτε να πληρώνουν τα σπασμένα, να πληρώνουν το τίμημα. Θα πρέπει να γίνουμε παγκόσμιοι ηγέτες αλλά να προσετεριστούμε και άλλου εταίρους και να επιδιώξουμε παγκόσμια υποστήριξη. Επίσης θα πρέπει να κινηθούμε νυφάλια και σοφά και συνετά. Να προωθήσουμε την κλιματική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια και να χρησιμοποιήσουμε και τους πολιτικούς μας φίλους και εταίρους προκειμένου να αισθενιστούν τη γνώμη μας παγκοσμίω. Ευχαριστώ και το λόγο έχει συνάδελφος η Μέρντ Μαγκίνες. Θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στους ομιλητές μας να απαντήσουν. Και είναι ενδιαφέρον ότι η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι αυτή. Μπορούμε να τα έχουμε όλα, να συγκεράσουμε κλίμα και προσδοκίες της κοινωνίας. Και αυτό το ερώτημα βεβαίως δεν, μπορώ, δεν μπορώ να το απαντήσω σήμερα. Είναι ένα εξαιρετικά πιεστικό ερώτημα. Και άλλοι ρώτησαν, η πολιτική είναι έτοιμη για αυτήν την εποχή. Δεν ξέρω αν τα μέλη του πάνελ θέλουν να απαντήσουν. Αλλά φαντάζομαι κάτι θα έχουν να παρατηρήσουν. Και το σίγουρο είναι μάλλον ότι όλοι θέλουμε. Μπορούμε όμως. Είναι καλό που βρισκόμαστε εδώ πάντω, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια, για να κάνουμε το επόμενο βήμα μαζί προς τα εμπρός. Λοιπόν, ποιος θέλει τον λόγο σου να αρχίσω ανάποδα από την κυρία Ναβάρο αυτή τη φορά. Ναβάρο, να εστιάσω στο τελευταίο ερώτημα. Στη νέα δυνατή μας πολιτική που προκρίναμε τον Δεκέμβριο αποφασίσαμε να μην χρηματοδοτήσουμε πλέον έργα φυσικού αερίου μετά το 2021. Θα επικεντρωθούμε λοιπόν σε ενεργειακά έργα τα οποία θα υποστηρίζουν, θα κρατήνουν στην απομείωση του ρόλου του άνθρακα στην οικονομία μας. Θα υπόψη μας όπως είπα τα έργα, τα ενεργειακά έργα τα οποία υποστηρίζουν την αποστασιοποίηση από τον άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει σαφεί πολιτικές, έχει τι δικέ πολιτικέ, πολιτικές, αλλά και εσεί ε, επηρεάζετε την πολιτική μας. Θα μας πείτε και εσείς τι πρέπει να κάνουμε και οι επιστήμονε μας θα μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Και ξέρουμε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, θα υπάρχει κόστος. Αν τα δούμε όμω τα πράγματα πιο μακροπρόθεσμα, τώρα συνειδητοποιούμε ότι Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε για το μέλλον των κοινωνιών μας και τον πλανήτη. Ευχαριστώ. Κύριος Ράιντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ενθερρυντική η συζήτηση. Ε, νιώθω ήδη πολύ αισιόδοξο. Δεν θα ήθελα να μας πάρουν από κάτω οι αρνητικές σκέψεις. Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι σωστός. Δηλαδή, οι φιλόδοξοι στόχοι μας είναι σωστοί και μπορούμε να τους πετύχουμε. Σαφώς μπορούμε. Οπότε ας μην ε, αφιερώσουμε τόσο πολύ χρόνο σε τεχνητά διλήμματα μεταξύ πλανήτη και θέσεων εργασίας. Κοιτάξτε, η μετάβαση αυτή πιθανότερα δεν έχει προηγούμενο σε αυτήν την κλίμακα τουλάχιστον και δεν θα είναι εύκολο. Ε, το είπε και ο Ρουμάνο συνάδελφο. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα. Η μετάβαση έχει τώρα κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ε, πρώτον, δεν είναι μια ελεύθερη επιλογή. Γίνεται υποπίεση. Ο πλανήτης στέλνει κραυγή αγωνίας. Και να μην ξεχνούμε επίση ότι η μετάβαση αυτή συμπίπτει χρονικά με άλλες μεγάλες μεταβάσεις της κοινωνίας μας. Την ψηφιακή μετάβαση, την δημογραφική μετάβαση. Γιατί ωραία τα λόγια, καλ... είναι ωραία η μετάβαση από τον άνθρακα στην ε, υψηλή τεχνολογία, αλλά έχουμε εδώ να κάνουμε με πολυάριθμες μεταβάσεις. Βέβαια, το καλό είναι ότι μπορεί η μία να βοηθάει την άλλη, να μην είναι αντιφατικές. Και ένα πολύ γενικότερο σχόλιο, που είναι και υποχρέωσή μου. Ε, τι γίνεται με τις ΗΠΑ και τι γίνεται με τις άλλες χώρες που δεν μας παίζουν. Αυτό είναι το μειονέκτημα για την Ευρώπη. Και όπως είπε και ο κύριος Μιλόσεβιτς, ε, χρειαζόμαστε να πάρουμε με το μέρος μας και τις ΗΠΑ. Αλλά υπάρχει και ο υπόλοιπο κόσμος που ζητά βοήθεια από την Ευρώπη σήμερα. Γιατί μπορούμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν και τη δική τους μετάβαση. Υπάρχουν χώρες, ξέρετε, που δεν έχουν τα εφόδια που έχουμε εμείς, δεν έχουν τη γνώση που έχουμε εμείς, που έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Να μην ξεχνούμε λοιπόν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλες χώρες οι οποίες δεν θέλουν να μείνουν πίσω. Ευχαριστώ και ο κύριος Καρνή. Ευχαριστώ. Τρία πράγματα. Να συγκεκριμένο ερώτημα αφορούσε την TCFD. Ε, ο κόσμος είπε κάποιος δεν ξέρουν τι είναι. Οι επιχειρήσεις, να σας διαβεβαιώσω, ξέρουν. Οι μεγάλε επιχειρήσει ξέρουν. Χίλιες ήδη μεγάλε επιχειρήσεις και κρατικές επιχειρήσεις που εκπροσωπούν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια υπέγραψαν και αποδέχτηκαν την υποχρέωσή τους να δημοσιεύουν στοιχεία που αφορούν το κλίμα. Μπορεί να μην έχει φτάσει ακόμη όντω ναι, στι μικρέ επιχειρήσει. Όμω ή τη σκεφτεί, θεσπίζει διαδικασίες, τις εφαρμόζει. Διαμορφώνει πολιτική. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία λοιπόν δημοσιοποίηση και μη χρηματοπιστωτικής φύσης στοιχείων, πολύ σημαντικό και είναι στα χέρια σας από εδώ και πέρα να το κάνετε να λειτουργήσει. Όμως, εδώ βρίσκεται η απάντηση του ιδρυτικού τομέα. Τι θα κάνει ο ιδρυτικό τομέα βάσει αυτών που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλέ άλλε χώρε. Στην πορεία προ το ουδέτερο ισοζυγείο. Δεύτερον, όσον αφορά τι κεντρικέ τράπεζε και το κατά πόσον παίζουν το παιχνίδι ή όχι, έχουμε 50 κεντρικέ τράπεζε μαζί με την τράπεζα της Αγγλίας έχουμε την Κινέζικη Τράπεζα και το καθεξής. Είμαστε πολλοί και ασχολούμαστε με τη διαχείριση κινδύνου. Και ο μεγαλύτερο κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, και αυτό το γνωρίζουμε από την εποχή τη κρίση, είναι μια ξαφνική κατάρρευση. Αυτόν τον κίνδυνο μειώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν οικονομικέ ευκαιρίε λοιπόν και έχουμε μπροστά μα, εγώ πιστεύω, μια τεράστια οικονομική ευκαιρία χωρίς να υποτιμούμε φυσικά το κόστος. Και πολύ γρήγορα, οι άλλα δύο σημεία. Ακούσαμε κάτι για τις ΗΠΑ, πολύ σημαντικός παράγοντας. Δεν συμμετέχει στην ΕΚΟΠ, τι θα γίνει με την ανταγωνιστικότητα των άλλων οικονομιών κλπ. Η ερώτηση είναι, η Αμερική θα παραμείνει για πάντα εκτός ΚΟΠ ή οι αμερικανικές βιομηχανίες έχουν διαφορετική γνώμη. Εγώ πιστεύω ότι και η καινοτομία σε πολύ μεγάλο βαθμό προέρχεται από την Ευρώπη, όχι επειδή γεννιέται εδώ αναγκαστικά, αλλά ε, γιατί έχουμε ευρωπαϊκέ εταιρείε που είναι παγκόσμιε, πολυεθνικέ. Αλλά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ειδικού τομεί συγκεκριμένα. Ας πούμε στην Ιταλία μιλούσαμε με έναν ειδικό για το μεθάνιο. Νομίζω ότι η Ιταλία ασχολείται περισσότερο με το φυσικό αέριο. Αλλά η Ιταλία είναι μπροστά σε αυτόν τον ε, τομέα. Η βιομηχανία του υδρογόνου θα μας βοηθήσει να συλλέξουμε διοξίδιο του άνθρακα. Είναι ένα τομέα στον οποίο ε, είμαστε πρωτοπόροι και έχουμε πολλές ευκαιρίε Λοιπόν, πιστεύω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ίσως θα θελήσουν να ακολουθήσουν στον δρόμο που χαράσουμε και έχουμε ευκαιρίε εξαγωγή τεχνολογία εκεί. Και για να κλείσω όσον αφορά την ανάπτυξη και την στάση της πολιτικής. Δεν είναι ανάπτυξη αν δεν είναι αηφορική. Αυτό το μάθαμε με την κρίση. Χρειάστηκε μια δεκαετία για να μάθουμε το μάθημά μας, για να βγούμε από το λάκκο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθυστερήσουμε την μετάβαση. σα ίσα χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα. Όπω είπε όμω και ο έστενο συναδελφό που μα προειδοποίησε, δεν αρκεί να εξηγούμε απλώ. Πρέπει ο κόσμο να καταλάβει γιατί πράγμα μιλάμε. Πρέπει να συμμετάσχει στην προσπάθεια. Ο κάθε ένα από εμά ξεχωριστά, στη βάση. Και αυτό είναι μέρος της πρόσκλησης πρόκλησης για την πολιτική και τους πολιτικούς. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι έχουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο, ότι έχουμε πρόγραμμα και αυτό πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένε δράσεις οι οποίες να, με τις οποίες να ταυτιστεί ο κόσμος, να νιώθει καλά αυτό το πρόγραμμα και εσείς ως κοινοβουλευτικοί το γνωρίζετε αλλά πρέπει να πείσουμε και ένα σωρό άλλες ομάδες που περιμένουν από εμάς να λύσουμε αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Πρέπει και αυτούς να φέρουμε στο πλευρό μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους σας ε, για τις ε, παρεμβάσεις. Ε, κοίταγα λιγάκι στο θεωρείο και εκεί βλέπω πάρα πολλούς νέους. Αυτή είναι και το μέλλον. Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει κάποιος ε, που θα θέλει να κάνει μια ερώτηση. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να ε, σηκώσετε το χέρι σας. Αν όχι, θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ εγώ. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ελέγχθησαν πολλά και σημαντικά. Ε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά το να το κάνει κανείς στην πράξη, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από το να το λέει. Θα καταλάβετε ότι εγώ έρχομαι από την Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία, κατά το παρελθόν, υπήρχαν αγροί με τύρφοι ε, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας ε, και τώρα σκεπτόμαστε να το σταματήσουμε αυτό. Ε, και όπως είπε και ο κύριος Μακάνη, το τοπικό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν δεν συμμετέχουν οι πολίτες επιτόπου τότε προκύπτουν διαμαρτυρίες οι οποίες ε, καθυστερούν ε, την ανάπτυξη. Νομίζω λοιπόν ότι όσον αφορά τα θέματα της πολιτικής, το συζητήσαμε με τον Συμπρόεδρο, πρέπει να έχουμε πολιτικές και λειτουργίες κάτω από αυτή τη νέα δυναμική. Γιατί εμείς λειτουργούμε στο πλαίσιο ενός πολιτικού κύκλου που είναι κάποια χρόνια αλλά αυτά είναι θέματα που μας ξεπερνάνε. Είναι πολύ πιο μακροχρόνια. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο στο πλαίσιο μιας έντονης ε, βραχυπρόθεσμης πολιτικής να μιλάει κανείς για τα μακροπρόθεσμα που μπορεί να είναι και πόδινα. Ε, ξέρω ότι ε, καθηγητές πολιτικής ε, έχουν ε, εξετάσει τα θέματα, το πώς λειτουργούμε. Βεβαίως καμιά φορά αυτό να είναι πολύ πιο εύκολο για έναν κεντρικό τραπεζίτη. Όμως η πολιτική ξέρετε εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα γιατί υπάρχει και κατακαιρματισμός. Οι άνθρωποι ψηφίζουν με διαφορετικούς τρόπους και μετά αναζητούν τη συνένεση. Εδώ ε, στο κοινοβούλιο που βρισκόμαστε εδώ είναι η καρδιά της συνένεσης έτσι ώστε κανείς να μην χάσει. Αυτή λοιπόν η συζήτηση για μια άλλη μέρα. Νομίζω ότι αναφέρθηκε η Γεωργία που είναι πολύ σημαντική για μένα. Η Γεωργία πράγματι χρειάζεται τη μετάβαση αλλά ξέρω επίσης ε, ότι οι Γεωργοί αυτή τη στιγμή αισθάνονται στοχευμένοι, ότι βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Ε, πρέπει όμως να τους πάρουμε με το μέρος μας ε, να ε, προχωρήσουμε από κοινού όσοι βρισκόμαστε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και νομίζω όλα αυτά έχουν σχέση και με τη βιομηχανία. Συνάδελφος από την Πολωνία είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τη συζήτηση την βρήκα πολύ σημαντική γιατί η δική μου ευθύνη είναι να ε, καλλιεργώ το διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και το λέω αυτό συνεχώς ότι πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα. Σήμερα είχαμε ένα πολύ καλό παράδειγμα που μπορέσαμε να ανταλλάξουμε απόψει για κάτι που αφορά όλους μας, είναι στην καρδιά μας ανεξάρτητα από την πολιτική μας τοποθέτηση. Πρόκειται για την μοίρα μας κοινή πολιτική στόχη Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται καλά τα πήγαμε με το χρόνο και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που έχουμε κοντά μας τον Επίτροπο ε, δεν ξέρω αν θα κάτσει το βήμα θα ήθελα τώρα να καλέσω τον κύριο Ντομπρόφσκη, ο οποίο είναι εκτελεστικό αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μα ε, μιλήσει για το πρόγραμμα επενδύσεων, τη ε, βιώσιμο πρόγραμμα επενδύσεων στην Ευρώπη. Και αν και πρέπει να φύγετε, μπορείτε να φύγετε, αλλά ε, να καλέσουμε τον Επίτροπο στο βήμα και βεβαίως να χειροκροτήσουμε πριν φύγουν τους ομιλητές μας. Είχαμε ένα μικρό διάλειμμα για τους φωτογράφους. Ε, χαιρόμαστε που είσαστε κοντά μας. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ε, κλιματική αλλαγή ε, και θα ήθελα τώρα να σας δώσω το λόγο για την ομιλία σας. Uh, uh, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πριν από ένα μήνα είχα έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρουσιάσω τον επενδυτικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ, αυτή τη φορά όμως παρουσία και των εθνικών βουλευτών. Σήμερα η κλιματική αλλαγή είναι ύψη προτεραιότητα και πρωταρχική ανησυχία των πολιτών. Και ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι ε, των Ευρωπαίων πολιτών ε, είχατε κέριο ρόλο στην ε, διατύπωση αυτών των ανησυχιών και την ανάδειξή τους ως ύψητη προτεραιότητα. Θα διαδραματίσετε επίσης σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών. Με τον κάθε χρόνο που περνάει οι αποδείξεις για το ανέκτητη ανάγκη για το κλίμα είναι πια αδιάσυστες. Πριν από ένα μήνα η Παγκόσμια Μετεωρολογική Οργάνωση επιβεβαίωσε ότι το 2019 είναι η δεύτερη θερμότερη χρονιά στα στο ιστορικό και το Δεκέμβριο οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η Γρυλανδία ε, χάνει πάγο με εφταπλάσιους ρυθμούς από τη δεκαετία του 90. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η τάση και τον περασμένο μήνα είχαμε τον ε, θερμότερο Ιανουάριο στα καταγεγραμμένα χρονικά με βάση την ε, Εθνική Υπηρεσία Οκεανών και Ατμόσφαιρας και την περασμένη εβδομάδα στην Αντακτική είχαμε πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά στην ιστορία. Προεδρία. Οπότε έχουμε πολλά παρόμοια συμπεράσματα. Τα περισσότερα είναι πρόσφατα από αυτά που σα ανακοίνωσα, αλλά δεν μπορούμε να τα αγνοούμε και δείχνει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη τη δράση. Γι' αυτό και η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών είναι η προτεραιότητα της, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία. Η Πράσινη Συμφωνία αποδεικνύει την αποφασιστικότητα και δέσμευσή μα να γίνουμε ουδέτεροι κλιματικά ήπειρο μέχρι το 2050, κάτι που θα κατοχυρωθεί και στην πρώτη κλιματική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που προποθέτει πρωτοφανή εξυγχρονισμό και μετασχηματισμό. Ε, σε τεράστια κλίμακα. Θα χρειαστεί αναδιάρθρωση και βιομηχανική, βιομηχανικός μετασχηματισμός σε όλες τις χώρες και φυσικά θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τις παραδοσιακές τεχνολογίες και να υιοθετήσουμε μηδενικές ε, ως προς τον άνθρακα εναλλακτικέ λύσεις. Φυσικά για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας για το 2030 θα χρειαστούμε 260 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον σε αιτήσεις επενδύσεις και αν ε, ενισχύσουμε τις ε, φιλοδοξίες μας για περιορισμό των εκπομπών θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε με ακόμη πιο δαψιλή κονδύλια την πράσινη μετάβαση. Βέβαια το κόστος της ε, αδράνειας θα είναι ακόμη πιο υψηλό. Για να υλοποιήσουμε λοιπόν την Πράσινη Συμφωνία χρειαζόμαστε ένα εύρωστο χρηματοδοτικό πλαίσιο και γι' αυτό ε, και γι' αυτό και μάλλον παρουσιάσαμε και το επενδυτικό σχέδιο που θέτει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των επενδύσεών μας και μάλιστα συνδυάζει νέε πρωτοβουλίε πολιτική με υφιστάμενου μηχανισμού και σηματοδοτεί μια αλλαγή νοοτροπία. Με τη δική σα υποστήριξη του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα προ τι δημόσιε αρχέ, τι εταιρείε και του επενδυτέ, ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε πράσινα όταν λαμβάνουμε επενδυτικέ αποφάσει. Το επενδυτικό μα σχέδιο θα μα δώσει μια σημαντική χρηματοδοτική όθηση δημιουργώντα πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ για την επόμενη δεκαετία για τη χρηματοδότηση βιώσιμων σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Και γι' αυτό αφιερώνουμε το, τουλάχιστον το 25% των δαπανών μας στη στήριξη, στήριξη των κλιματικών αλλαγών. Και μάλιστα αυτό σε μία δεκαετία θα ανέλθει σε 503 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία μας μερίδιο δημόσιων κονδυλίων. Και επίσης ε, θα μοχλεύσει 114 δισεκατομμύρια ευρώ σε εθνική συγχρηματοδότηση για κλιματικά και περιβαλλοντικά σχέδια. Το επενδυτικό μας πρόγραμμα Invest EU θα επικεντρωθεί κυρίως στην βιωσιμότητα και θα μοχλεύσει περίπου 279 δισεκατομμύρια ε, δημόσια και ιδιωτικά κονδύλια για κλιματικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις μεταξύ 2021 και 2030. Από από το InvestEU ε, και με, την, ε, και με την εγγύηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για να προσελκύσουμε επενδυτές θα μπορούσαμε να επενδύσουμε και σε πιο ε, σημαντικά περιβαλλοντικά σχέδια και θα αξιοποιήσουμε τα δημόσια κονδύλια για το δημόσιο καλό. Και με την εγγύηση αυτή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορεί να επενδύει σε σχέδια υψηλότερου κινδύνου, κάτι που θα προσελκύσει και ιδιώτες επενδυτέ. Και πέραν του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε και το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ίσως της σημαντικότερης μετάβασης και του σημαντικότερου μετασχηματισμού σε αυτόν τον αιώνα και θα είναι εφικτός μόνο εφόσον είναι δίκαιος και λειτουργεί για όλους. Και αυτό είναι ο στόχος του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης που ε, θα παράσχει περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θα επικεντρωθεί σε ανθρώπους και περιοχές που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα ή από διαδικασίες έντασης άνθρακα σε κατοίκους περιοχών που εξαρτώνται από τον άνθρακα για παράδειγμα και βρίσκονται σε μετάβαση. Επίσης θα στηρίξει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, την διαφοροποίηση και τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό οπότε να ξαναβρούν δουλειά στην αγορά εργασίας οι πολίτες που την έχουν χάσει. Επίσης θα έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες ε, της μετάβασης. Όλα αυτά θα συζητηθούν ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ενδιαφερομένων χωρών. Βέβαια, ο μηχανισμός δικής μετάβασης δεν αφορά μόνο δεξιότητες και χρήματα. Θα παράσχει και τεχνική υποστήριξη σε κράτη-μέλη και επενδύσεις, κυρίως στις πληγήσεις περιοχές, στη τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς εταίρους και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Επίσης είναι και η υπόσχεσή μας ε, για την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι θα με υποστηρίξετε και εσείς από το Κοινοβούλιο και τα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό αυτή την πρωτοβουλία. Και φυσικά ε, με τα δημόσια κονδύλια δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το σύνολο της πράσινης μετάβασης. Θα πρέπει ε, να προσελκύσουμε και ιδιωτικά κονδύλια. Και σίγουρα τα δημόσια κονδύλια θα χαράξουν το δρόμο, αλλά ο ιδιωτικός κλάδος θα εξασφαλίσει οικονομία κλίμακος. Και με ε, στοιχεία του ενεργητικού πάνω από 100 εκατομμύρια. ο χρηματοπιστωτικό ε, κλάδο έχει τεράστιο δυναμικό για, πράσινες, για πράσινε επενδύσει. Και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπω τράπεζε, ασφαλιστικέ εταιρείε, ε, συνταξιοδοτικά ταμεία και επενδυτικά ταμεία θα πρέπει να βρουν τα σωστά εργαλεία για να επενδύσουν πράσινα. Και με την ταξινομία ε, θα επιλέξουμε τις δραστηριότητες που θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμες για να επενδύσουμε. Και φυσικά τώρα που έχουμε τις βασικές αρχές θα πρέπει να ε, θέσουμε σε ισχύ το σύστημα. Και χαίρομαι που πριν την έναρξη ακόμη ισχύω, ήδη κάποιες εταιρείε χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα για να ε, κάνουν μια βολιδοσκόπηση ε, και φυσικά θα έχουμε με την ολοκλήρωση της ταξινομίας το πράσινο ομόλογο και το, την οικολογική σήμανση. Μάλιστα, στη συνέχεια του έτους σας παρουσιάσουμε την ανανεωμένη στρατηγική για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά. Και φυσικά θέλουμε ε, δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών ε, πληροφοριών από τις εταιρείες. Είναι ε, σημαντικά αυτά τα πρότυπα και θα βοηθήσουμε έτσι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, θεσπίσει κάποιες πανευρωπαϊκές ε, προδιαγραφές για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. Έτσι θα έχουμε πρότυπα και σήματα για βιώσιμα προϊόντα και επενδύσεις. Και βέβαια ένα θέμα είναι να έχουμε τη σωστή χρηματοδότηση και άλλο να έχουμε τη σωστή πολιτική και το κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό είναι σημαντικό για να καθοδηγήσουμε τους επενδυτές προς βιώσιμες επενδύσεις και να καθοδηγήσουμε τις αλλαγές στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Για παράδειγμα, θα προτείνουμε κανόνες για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι το 2021 θέλουμε να προσαρμόσουμε τους κανόνες μας για κριτικές ενισχύσεις ώστε να αντικατοπτρίζουν τους στόχους της πράσινης συμφωνίας και στο δημόσιο τομέα συνεργαζόμαστε με, πράσινε, με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να δημιουργήσουμε κριτήρια αναφοράς για τις δημοσιονομικές πρακτικές. Και για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα, θα περιλάβουμε και το κριτήριο της βιωσιμότητας της αναχώρα εκθέσεις. Ε, θεωρώ το επενδυτικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας ε, ως σημαντικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση του ευρύτερου αγώνα μας στην Ευρώπη για τις κλιματικές αλλαγές. Και η, στρατηγική μας θα οδηγήσει σε έναν ρηξικέλευθο μετασχηματισμό, θα προστατεύσει το περιβάλλον, θα εξυγχρονίσει την οικονομία για ένα βιώσιμο μέλλον, θα αυξήσει τις επενδύσεις ε, σε πιο ε, ανταγωνιστικές τεχνολογίες και θα εξασφαλίσει καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Όσο περισσότερο επικεντρώσουμε, συγκεντρώσουμε χρηματοοικονομικές ροές, τόσο περισσότερες θέσεις απασχόλησης θα προστατεύσουμε και θα προασπίσουμε και το περιβάλλον και το φυσικό μας κόσμο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την προσοχή σας, αλλά και για την υποστήριξή σας στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ για την λεπτομερή ανάλυση της επενδυτικής μας στρατηγικής και τώρα ο λόγος στον κύριο Μίχελ Πάχ από την Γερμανική Βουλή που έχει μια πρόσκληση να μας απευθύνει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία εκ μέρους του συνόλου της ε, γερμανικής αντιπροσωπείας από το Bundestag να σας προσκαλέσω στο Βερολίνο στην επόμενη συνεδρίαση σε μια διάσκεψη η οποία θα λάβει χώρα 12 και 13 Οκτωβρίου του 2020 στο Reichstag του Bundestag. Και αυτή τη στιγμή ε, προετοιμάζουμε για σας ένα πολύ ελκυστικό πρόγραμμα για να συζητήσουμε τα επίκαιρα θέματα, ε, πολύ ενδιαφέρουσες οι προσωπικότητες που έχουμε προσκαλέσει και ελπίζουμε κυρίως ε, η προερχόμενη από τη Γερμανία, κυρία Φονταλάι, να είναι και αυτή παρούσα. Προσβλέπουμε σε μια ζωντανή ανταλλαγή απόψεων με όλους σας και χαιρόμεθα που μπορούμε να σας προσκαλέσουμε ή θα χαρούμε πολύ να σας δεχτούμε στο Βερολίνο να είστε όλοι υγιείς και χαρούμενοι. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πω αντίο και προσβλέπουμε στο να σας δούμε στο Βερολίνο. Πρόεδρος. Σήμερα το πρωί τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά ε, με τις ομιλίες. 12 και 20 θα ξανάρθει ο κύριος Σασόλη για την οικογενειακή φωτογραφία. Θα έλεγα λοιπόν να έρθετε και πάλι πίσω στις 12 και 20 και μετά θα ακολουθήσει το γεύμα. Αλλά προς το παρόν διάλειμμα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για τις παρεμβάσεις σας. Ήταν όλα ιδιαίτερα κατατοπιστικά. Ε, σύντομο διάλειμμα λοιπόν.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 can he be seated, seated or, or he be seated, or standing up? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Παρακαλώ προχωρήστε για τη φωτογραφία, για την ομαδική φωτογραφία. Ελάτε στις πρώτες σειρές παρακαλώ να μαζευτούμε για να βγάλουμε την ομαδική φωτογραφία. The picture will be taken like this. From here. From here. Standing up. Or... And φωτογραφία θα ληφθεί από το Προεδρείο. Γι' αυτό πρέπει να είστε κοντά. Παρακαλούμε, πλησιάστε. To them, they will help you. The speaker in the front. And the speaker in the front, please.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 Dear colleagues, dear colleagues, perhaps the most important announcement or reminder is that lunch will be served in one minute or two, and it is. Η πιο σημαντική ανακοίνωση. Σε ένα-δύο λεπτά θα αρχίσει το γεύμα στον πρώτο όροφο στην αίθουσα, το χώρο τέλος πάντων, για Χούντι Μενουχίν.